Mm, παρακαλώ, καθίστε συνάδελφοι. Μπορούμε να αρχίσουμε με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σας παρακαλώ να καθίσετε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε με τις εργασίες μας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Νίκολα Γκαμπούρο, Γενικό Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και θα είναι σε επαφή μαζί μας μέσα στα πλαίσια των νέων του καθηκόντων επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μαρόκο. Γιατί όπως ξέρετε το Μαρόκο βρίσκεται σε εταιρική σχέση, ενισχυμένη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο κύριος Λανταμπούρου, ο Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων, θα ασχοληθεί και με το θέμα του Μαρόκου, την εταιρική σχέση. Σήμερα βρίσκεται εδώ υπό μία συγκεκριμένη ιδιότητα. Θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις της ενεργειακής ασφάλειας μετά από την υπογραφή της 13ης Ιουλίου για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και θα μας μιλήσει και για άλλα θέματα μεταφοράς ενεργείας μέσα στα πλαίσια του διαδρόμου του Νότου. Υπάρχει και το South Stream, όπως ε, γνωρίζετε, που θεωρείται από τη χώρα μου και από άλλες χώρες ε, ένα ανταγωνιστικό σχέδιο σε σχέση με τον Ναμπούκο. Το κοινοβούλιο μας αποφάσισε να προωθήσει μία συζήτηση κατά την επόμενη Ολομέλεια και έτσι εμείς θα προβούμε στην ε, προετοιμασία αυτής της συζήτησης. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να λάβουν υπόψη ότι μπορεί να προβάλλουμε μία προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συζήτηση στα μέσα του Σεπτεμβρίου σε σχέση με τις επιπτώσεις της εξωτερικής πολιτικής στον ε, ενεργειακό τομέα. Αυτό το προσχέδιο προφορικής ερώτησης που έχει οριστεί από τους συντονιστές θα σας διανεμηθεί και έτσι θα μπορέσετε να σχολιάσετε και ενδεχομένως να αλλάξετε κάπως την προφορική ερώτηση. Μετά την ε, παρέμβαση του κυρίου Λανταπούρου δεν είναι ακόμα μαζί μας, αλλά προτρέχω κάπως. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάριος ε, Βόλσκι, ο οποίος ήταν και προκάτοχος του αξιώματός μου και όπως ξέρετε ασχολήθηκε με ενεργειακά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι ο φυσικός μας εκπρόσωπος επί του θέματος και θα ακούσουμε και τη δική του γνωμοδότηση πριν ανοίξει η συζήτηση. Δεν έχω άλλα σχόλια επί του παρόντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λανταμπούρου και του δίνω το λόγο θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ όλους για την εκλογή σας στο αξίωμα αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μελλοντικά σας καθήκοντα είναι ολοένα και μεγαλύτερα τη στιγμή που θα πρέπει να ορίσουμε μια εξωτερική πολιτική, μια δυνατή εξωτερική πολιτική, εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Ελπίζω να κυρωθεί και η συνθήκη της Λισαβόνας και όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική σας Επιτροπή θα φέρει μεγάλες ευθύνες και αρμοδιότητες για την εφαρμογή των συνθήκων και συγκεκριμένα τις συνθήκες της Λισαβόνας που διανοίγει μεγάλες δυνατότητες για να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε γενικότερα μια κοινή εξωτερική πολιτική. Σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω να συνεισφέρετε στο στο ευρωπαϊκό ζήτημα και οικοδόμημα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ιδιαίτερα γιατί θα σας αναπτύξω αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Έξι χρόνια είμαι Γενικός ε, Διευθυντής των Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής και με απασχόλησε αυτό το ζήτημα το οποίο κατέχει όλο ένα και σημαντικότερη θέση στο παγκόσμιο σενάριο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Όλοι θα θυμόσαστε τα γεγονότα που ε, αντιμετωπίσαμε με την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να, μας, να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας με ολέθριες συνέπειες για ορισμένα από τα κράτη-μέλη μας. Αυτό αποτέλεσε πραγματικότητα. Θα θυμόσαστε ότι εδώ και ένα χρόνο στην κρίση, κατά την κρίση της γεωργίας υπήρξαν δραματικές επιπτώσεις ως προς την κυκλοφορία και προμήθεια, ενεργειακή προμήθεια σε, ε, στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου υπάρχουν γεωπολιτικές ανησυχίες, υπάρχουν κλειδονισμοί ε, των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό έχει επιπτώσει συλλογικά και ατομικά στα κράτη-μέλη. Το κεντρικό θέμα αφορά τη συλλογιστική μας σε σχέση με το ρόλο της Ευρώπης ως προς τις εθνικές πολιτικές που στιγματίζουν την ε, γεωπολιτική μας πραγματικότητα ως προς την ενεργειακή ασφάλεια. Και η Επίτροπη με μετριοφροσύνη χρησιμοποιώντας τις αρμοδιότητες της παρούσης συνθήκης προσπάθησε να προκαλέσει μια συζήτηση στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να μιλάμε με μία φωνή. Φέρω την ευθύνη να είμαι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τη ρωσική κυβέρνηση για να φτάσουμε σε μία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν ε, βρεθώ στη Μόσχα, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με μία φωνή, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες ε, από όταν μιλάμε μεμονωμένα και κατακαιρματισμένα. Αυτές είναι οι προθέσεις μας, χωρίς να το επιτυγχάνουμε πάντα. Δεν έχουμε αυτή την κοινή θέση που μας δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες ε, παρέμβασης. Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, αποφασίσαμε και επιτύχαμε το εξής. Η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο, στην υψηλότερη βαθμίδα των διμερών σχέσεων που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Είχα συμμετάσχει σε όλες τις διασκέψεις κορυφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις κυριότερες χώρες και αυτό το ζήτημα το, το θέτουμε σε κάθε περίσταση. Το θίξαμε με τις ΙΠΑ, με τη Μόσχα, με την Κίνα, με την Ιαπωνία, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και με όλες τις ε, χώρες γενικότερα του Μερκοσούρ. Είναι ένα κατά προτεραιότητα θέμα ως προς τις διεθνείς σχέσεις. Επίσης, προσπαθήσαμε και καταφέραμε εμπολής να συζητήσουμε με τους εξωτερικούς εταίρους για το ευρωπαϊκό ενεργειακό πρότυπο ως προς την κυκλοφορία και προμήθεια σε ενεργειακά προϊόντα και αυτό μας ε, οδηγεί στο να επηρεάζουμε την κατάσταση σε σχέση με την ε, Λατινική Αμερική και τις χώρες ΑΣΕΑΝ διότι όλες οι χώρες προβαίνουν σε μια περιφερειακή ολοκλήρωση μέσα στα πλαίσια των ε, αγαθών και προϊόντων. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πω ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο σύγκρισης. Επίσης, θέσαμε σε εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις ενεργειακές κρίσεις καλύτερα. Μάθαμε από το μεγάλο μάθημα της Ουκρανίας και τώρα διαθέτουμε ορισμένους μηχανισμούς διάθεση πληροφοριών και ανταλλαγής πληροφοριών και μηχανισμούς ε, ανταπόκριση στην ε, κρίση που δεν υπήρχαν ε, εδώ και λίγους μήνες. Τώρα υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ενσωματώσαμε το θέμα της ενέργειας στην γεωπολιτική μας στρατηγική ασφάλειας. Ξέρετε ότι τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε με τον Χαβιέ Σολάνα, με τον ύπατο εκπρόσωπο, ως προς την επικαιροποίηση, με την επικαιροποίηση μάλλον της στρατηγικής μας σε θέματα ασφάλειας. Και δεν χωρεί αμφιβολία ότι το 2003 με βάση τις εξελίξεις που είχαμε καταφέραμε να ενσωματώσουμε σε αυτές τις προτεραιότητες ευρωπαϊκής ασφάλειας και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Υπάρχει και το δίκτυο των ανταποκριτών στην ενεργειακή ασφάλεια που ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα πρέπει να τονίσω ότι ε, θέλουμε την υποστήριξη της δικής σας Επιτροπής. Μιλήσατε για τις ε, εργασίες του Σάριους Βόλσκι στην, ε, παλαιά, ε, στην προγενέστερη Επίτροπη, ο οποίος συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε επί μιας κοινή θέσης με κέρυες αποχρώσεις ίσως αλλά ο κύριος Πέτεριν επίσης μας βοήθησε και ενίσχυσε αυτή την πρόταση πολιτικής υφής. Η Επιτροπή αυτή υπό την αιγίδα του Σάριους Βόλσκι συζήτησε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται ή άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Θα υπάρξουν εξελίξεις, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική πρόταση η οποία θα συζητηθεί και στο μέλλον. Με λίγα και απλά λόγια. Καταφέραμε μερικά χρήσιμα πράγματα, όμως η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Είμαστε πεπισμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για να μπορέσουμε να δράσουμε και για να μπορέσει να έχει επιρροή η Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγαλύτερο βήμα στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό τομέα. Το είπα κατά την εισαγωγή μου και αυτό θα είναι και, αυτή θα είναι και η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος. Εάν κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι, θεωρώ ότι ε, διανοίγει νέες δυνατότητες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγαλύτερες και περισσότερες αρμοδιότητες για την καλύτερη εργασία της και για την κατάρτιση μιας στρατηγικής και δυνατότητας θέσης σε ισχύ αυτής της στρατηγικής. Αυτό είναι το βασικό καθήκον της ε, Μελλοντικής Επιτροπής και ελπίζω να μην αρκεστούμε στην ε, στρατηγική, μέχρι τούδε στρατηγική δηλαδή να μιλάμε με μία φωνή, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο αλλά όχι επαρκές, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε καλύτερη εταιρική σχέση με τους ε, εταίρους μας γενικότερα. Επειδή θα βρίσκομαι για τελευταία φορά σε αυτή την Επιτροπή, θα ήθελα να λάβετε υπόψη την εξή σκέψη για το μέλλον. Δεν πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αρκεί για να δώσει στην Ευρώπη τις δυνατότητες να ορίσει και να προωθήσει μια ενεργειακή πολιτική που να προβάλλει αποκλειστικά τα συμφέροντα της Ευρώπης. Υποστηρίζω την πρόταση του Ζακ Ντελό εδώ και 1,5 χρόνο στον γαλλικό τύπο που ζητούσε μία συνθήκη, μία συνθήκη μόνο για θέματα ενέργειας που να είναι ισόβαθμη της ΕΚΑΧ έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ε, αμοιβαίο σύστημα διανομής και προμήθειας, όπως ίσχυε με τον άνθρακα και τον χάλιβα. Θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να μοιραστούν αυτή την κυριαρχία έτσι ώστε να προβάλλουμε ένα δίκτυο αμοιβαιότητας για να έχουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Ξέρουμε πως έχει η κατάσταση με τη Ρωσία. Εξαρτόμαστε από τη Ρωσία για την παροχή φυσικού αερίου. Ο μόνος τρόπος για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και των πολιτών και της ενεργειακής ασφάλειας είναι να προβούμε σε αυτό τον μεγάλο συμβιβασμό με τα κράτη-μέλη. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω σε, για ορισμένα ζητήματα επικαιρότητας. Το θέμα της ε, κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, της έντασης αυτής οι Ρώσοι πολλές φορές είπαν ότι θα, θα κλείσουν την παροχή διότι η Ουκρανία έχει υψηλά χρέη και οφειλές σε σχέση με προγενέστερες προμήθειες. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αποτελεσματικά το, την προηγούμενη άνοιξη και το καλοκαίρι. Επειδή μας εμπιστεύτηκαν και οι δύο κυβερνήσεις, η Γενική μου Διεύθυνση διαπραγματεύτηκε με τους διάφορους φορείς, έτσι ώστε να μην διακοπεί η παροχή ενέργειας η παροχή φυσικού αερίου. Η Ουκρανία πρέπει να πληρώνει το φυσικό αέριο που προμηθεύεται από τη Ρωσία μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας που υποστηρίξαμε όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέτρεψε ώστε τα χρήματα που ε, δίδονται στην Ουκρανία να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να πληρώσει τα τιμολόγια της Ρωσίας. Κατά δεύτερο λόγο, χρειάστηκε να επιβάλλουμε μία εσωτερική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυγχρονίσει το σύστημα δικτύων αεριαγωγών, έτσι ώστε στην εθνική της νομοθεσία να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές για να είναι διαφανής η αγορά. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει αναλάβει τη σχετική δέσμευση και η BERD, η ΕΤΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα καταβάλουν τα, τις αναγκαίες πιστώσεις για τον ε, εξυγχρονισμό του δικτύου της Ουκρανίας. Υπάρχει ένταση και κανείς δεν ξέρει μέχρι πότε η Ουκρανία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ε, υποχρεώσεις της και δεν θα ανακύψει μία νέα κρίση που θα μας επαναφέρει στην κατάσταση μερικών μηνών πριν. Εν πάση περιπτώσει, διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και θα συνεχίσουμε να ε, κατέχουμε αυτό τον ηγετικό ρόλο. Ως προς τον διάλογο με τη Ρωσία, μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συμφωνίας ε, Πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ε, θέμα της ενέργειας βρίσκεται στην υψηλότερη βαθμίδα. Η θέση μας δεν είναι κοντινές, διότι η Ρωσία δεν θέλει να προσυπογράψει, να κυρώσει μάλλον την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Χάρτα και ο πρόεδρος Μετβέντεφ ε, προέβαλε μία εναλλακτική λύση που δεν μας πείθει, διότι δεν αποτελεί επαρκή δέσμευση, έτσι ώστε η Ρωσία να δράσει σωστά ως προς την ε, διάβια, τη διαφάνεια μάλλον και την συνεργασία που θα πρέπει να προβληθεί. Μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες αν θέλετε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Σε αυτή τη συμφωνία με τη Ρωσία, στο τέλος θέλουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία ενεργειακής ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας ως προς τις ποσότητες και τους όρους παροχής τους όρους προμήθειας. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το επιτύχουμε αυτό, γι' αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και η δική σας Επιτροπή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το θέμα του νότιου διαδρόμου στην Πράγα είχαμε μία συνάντηση την Άνοιξη έτσι ώστε να διευρύνουμε τις δυνατότητες παροχής ενέργειας από όλες αυτές τις ε, χώρες του Νοτίου Καυκάσου δηλαδή και από πλευράς ε, Ιράκ, Ιράν και Αιγύπτου. Μπορούμε να επεκταθούμε επί του θέματος, αλλά είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Για ποιο λόγο. Θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε επαρκείς προμήθειες από τη Ρωσία. Η στρατηγική μας είναι να μειώσουμε αυτή την, ε, την παροχή, μάλλον αυτή την εξάρτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών πηγών, αλλά πρέπει να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση διανοίγοντας νέες αγορές με όλο το Νότιο, και, Νότιο Κάφκασο και την Κεντρική Ασία που θα μπορούσαν να είναι προμηθευτές φυσικού αερίου είναι το θέμα του Ναμπούκο που αναφέρθηκα, στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο μας απασχολεί. Προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτές τις δυνατότητες αγοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, ακόμα και από την Αλγερία και από άλλες χώρες. Αυτά θα είναι τα σημαντικά ζητήματα. Αν θέλετε θα μπορέσουμε να επεκταθούμε κατά τη συζήτηση. Ένα τελευταίο στοιχείο. Γνωρίζετε ότι πέρυσι προσπαθήσαμε να επανεκκινήσουμε την διαδικασία της Βαρκελόνης και τη Μεσογειακή Ένωση που ήταν μια πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας και ιδιαίτερα του Πρόεδρου Σαρκοζή, στα πλαίσια αυτής της επανεκκίνησης της Μεσογειακής Ένωσης, έχουμε ορισμένα προσχέδια ενεργειακής συνεργασίας και μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα σημαντικό σχέδιο που αφορά την πρόθεση της ηλιακής ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, θα αρκεστώ σε αυτά. Θα ήθελα να τονίσω τις ε, εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων και της ε, Επιτροπής σας. Όπως σας είπα, η συνθήκη της Λισαβόνας διανοίγει νέες δυνατότητες και η Επιτροπή σας θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ε, πολύ καλή πλαισίωση στα πλαίσια μιας μελλοντικής πιο ενισχυμένης συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Δόκτωρα Λάντεμπούρου. Στο μεταξύ βρίσκεται μαζί μας ο, προ, ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Πέτεριν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην πρόεδρος, και ο κύριος Σάριους Βόλσκι, ο οποίος ήταν εισηγητής ε, για θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας. Είναι ο φυσικός μας εκπρόσωπος επί των θεμάτων και του δίνω το λόγο. Θα ήθελα να σας πω εκ των προτέρων ότι έχουμε έναν κατάλογο 13 ομιλητών και πρέπει να ε, κλείσω τον κατάλογο. Διαφορετικά θα υπερβούμε κατά πολύ τον χρόνο μας. Ο κύριος Σάριος Βόλσκι έχει το λόγο. Uh, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αν εξετάσουμε πού βρισκόμασταν πριν από δύο-τρία χρόνια στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας μπορούμε με ικανοποίηση να ε, σημειώσουμε ότι έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδους και νομίζω ότι υπήρξε συνέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρισκόταν αρχικά ε, πολύ απασχολημένο λόγω ε, είχε ενδιαφερθεί για την ανάγκη να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα, καλή συνέργεια και με την Κομισιό που έχει τις δράσεις και τα έγγραφα και τα μέσα τα οποία αναφερθήκατε. Ε, έχουμε καταλάβει πολύ καλύτερα ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιό και παρατηρώ με ικανοποίηση ότι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την άποψη ότι μια ισχυρή φωνή ε, για την ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί ε, θεσμική διαρρύθμιση. Ε, στην έκθεσή μας προτείνουμε ε, και νομίζω ότι η μελλοντική ε, Κομισιόν θα έχει μια θέση η οποία θα είναι ισχυρότερη. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η συνθήκη, διότι πάντοτε αναφερόμεθα στη συνθήκη της Λισαβόνας ως ε, μια συνθήκη η οποία θα παρέχει καλύτερη νομική βάση για δράση. Αλλά ακούγοντά σας βλέπω ότι αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά αυτό είναι ένα θετικό σημείο από εμά, διότι θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο βάση της συνθήκης, με βάση τη συνθήκη και με τα όσα παρέχει, ούτω ώστε εμείς ε, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα μας. Και αυτό ισχύει επίσης με αυτό που είπατε, την πρόταση του Jacques Delors, ε, να έχουμε ε, να υπενθυμίσουμε τις αρχές που είχαμε, την κοινότητα άνθρακα και χάλιβα. Νομίζω ότι η νέα Κομισιόν, ε, θα δώσει ε, πολύ ε, καλύτερες και στερεές βάσεις στην ενεργειακή ασφάλεια λόγω της πείρας που έχουμε ως Ένωση, λόγω της άποψης της συμπεφωνημένης ότι πρέπει να μιλάμε με μία φωνή και να έχουμε μέσα και το βέλτιστο για μας θα είναι ε, να κοινοτικοποιήσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια. Ευχαριστώ την Κομισιό για την συνέργεια, τη συνεργασία μαζί μας με το Κοινοβούλιο και κυρίως ε, με αυτήν την Επιτροπή που θα έλεγα με κάθε μετριοφροσύνη ότι παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Και προσδοκούμε μελλοντική συνεργασία για την ανάπτυξη αυτής της εικόνας της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής στο μέλλον, πάνω σε όλες τις βάσεις, τις θεσμική, τα νομικά μέσα, ε, τα οικονομικά μέσα και ακόμα ε, και την παρακολούθηση αυτών των θεμάτων, ε, τις προτεραιότητες όπως τον Ναμπούκο <clears throat> που αναφέρατε και όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, είμαι αισιόδοξο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση είναι τελείως ικανοποιητική. Ποτέ δεν θα είναι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις και με τα νέα μέσα και τη νέα Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σάριους Βόλσκι και ξεκινάμε τη συζήτηση με την σύσταση, δυσάρεστη βέβαια, να αρκεστείτε σε 1,5 λεπτό. Ο κύριος Σαλαφράνκα, καταρχήν. Εντάχει κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να γενικό διευθυντή που βρίσκεται μαζί μας. Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας είναι ένα ε, θέμα φλέγων και εκρεμές και εδώ υπάρχει άμεση ανάγκη να επιλύσουμε τα ουσιαστικά ζήτηματα που απασχολούν τους ε, πολίτες μας. Γι' αυτό ο κύριος ε, Σάριος Βόλσκι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το τόνισε και ο κύριος Λανταμπούρου και θα πρέπει να εξέφρουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να επιβάλλει λύσεις σε αυτό το σοβαρό ζήτημα. Καθίσταται σαφές ότι ένα, ένας από τους τομείς αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις ως προς την ε, νέα συμφωνία με τη Ρωσία. Ποια είναι τα νέα στοιχεία και μηχανισμοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Λανταμπούρου φέρει μεγάλες ευθύνες και αρμοδιότερες ως ε, Γενικός Διευθυντής ε, Περιφερειακής Πολιτικής και στη συνέχεια υπεύθυνο διεύρυνσης. Τώρα είναι Γενικός Διευθυντής ε, Εξωτερικών Σχέσεων. Έχει έναν κατάλογο προτεραιοτήτων και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, όπως έκανε και υπό τις προηγούμενες ιδιότητές του. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσει να συνεισφέρει έμπρακτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις νέες του αρμοδιότητες και ελπίζω ο κύριος Λανταμπούρου να μπορέσει να παρευρεθεί και εδώ μέσα στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων του και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα, στην ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαφράνκα. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Πασκού για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Λανταμπούρο για την ε, παρουσίασή του. Αυτό μας δείχνει ότι αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα στο πρόγραμμά μας και θα εξακολουθήσει να είναι. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια αναπόφευκτα, τίνουμε να στρεφόμαστε προς τη Ρωσία, τόσο επειδή η Ρωσία είναι από τους βασικούς μας προμηθευτές, αλλά επειδή, ε, και, ε, επειδή παίζει ρόλο πολιτικό με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή της Επιτροπής πάνω στο ότι η ασφαλής ενέργεια δεν μιλάω για ενεργειακή ασφάλεια, αλλά για ασφαλή ενέργεια θα μπορούσε να επιτευχθεί εκτιμώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Και ξέρετε ότι οι μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, που παράγουν ενέργεια θα μπορούσαν με καλύτερο συντονισμό και καλύτερη σχέση θα μπορούσαν να δώσουν στην Ένωση ένα σημαντικό ποσοστό ασφαλούς ενέργειας. Και θα ήθελα τέλος να κάνω μια έκκληση ούτω ώστε ε, να αποδώσουμε σημασία και στην Ανατολή και στη Δύση, όχι μόνο στην Ανατολή όσον αφορά το θέμα της ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί τηρήσατε και το χρόνο. Ο συνάδελφος Βότσον για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα των φιλελευθέρων να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λανταμπούρο για την σημαντική εργασία που κάνει εξ ονόματο της Ένωσης ε, και για τις υπηρεσίες του μέχρι τώρα και να επαναλάβω την επιθυμία που εξέφρασε ο κύριος Σαλαφράνκα ότι στο ε, μέλλον ε, θα έχει μεγάλο βαθμό ικανοποίησης κύριε Πρόεδρε, κύριε Λανταμπούρο. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα μέσα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και θα μπορούσε να μας πληροφορήσει γι' αυτό ο κύριος Λανταμπούρο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η υπογραφή μεταξύ της Ρωσίας και τεσσάρων κρατών μελών της Συμφωνίας για τον αγωγό South, South Stream είναι το τελευταίο παράδειγμα του πόσο κατακερμακισμένη είναι η πολιτική μας ως προς την προμήθεια ενέργειας, τον εφοδιασμό ενέργειας. Μερικοί από εμά εδώ έχουμε έναν επικίνδυνο βαθμό ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία που θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει απειλή για την ακαιρεότητα της Ένωσής μας. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν ε, δύο ε, διέξοδοι ε, σε σχέση με αυτό το δίλημα. Να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην παραγωγή ενέργειας εντός των συνόρων μας. Έχουμε επίσης και την πυρηνική ε, ε, λύση που ευνοούν μερικοί και η άλλη λύση είναι οι μαζικές επενδύσεις σε ανανόσιμες πηγές ενέργειας και να βρούμε επίσης τους έξυπνους τρόπους για τους οποίους μίλησε ο κύριος Λανταμπούρο. Αναφέρθηκε σε αυτούς τους τρόπους όταν μίλησε για την ενδεχόμενη ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας σε συνεργασία Ποιο με τη Μεσόγειο. Ε, ποιος είναι ο βαθμός και η φύση των προσφάτων ε, συζητήσεων μεταξύ της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ρελέξ και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και ποιες είναι οι θέσεις οι σχετικές του Συμβουλίου για την ανάπτυξη μεγαλύτερου βαθμού αυτάρκειας ενεργειακής. Ευχαριστώ τον κύριο Βάτσον. Τώρα δίνω τον λόγο και σας παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο των 1,5 λεπτού ο κύριος Γκουτσκάφερ. Κύριε Γενική Διευθύντα, συγχαρητήρια για τη μελλοντική σας θέση και τη διπλωματική σας παρουσίαση. Συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Πρώτον, πιστεύετε ότι η συνύπαρξη, η αντιπαλότητα South Stream και Ναμπούκο μπορεί να αυξήσει την εξάρτηση της ε, Ευρώπης από την ενέργεια και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, τώρα ε, η Gazprom συμμετέχει κατά 50% σε, ε, μια, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και σε, κατά πόσο επηρεάζει αυτό το Ναμπούκο. Επίσης, το Economic Recovery Program ε, έγινε αναφορά και για την ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων η Κομισιόν έκανε μία μελέτη σε σχέση με την δυνατότητα υποστήριξης γειτονικών χωρών για να αυξήσουν την ε, ενεργειακή τους επάρκεια. Ε, ε, πώς θα προχωρήσει η Κομισιόν εδώ. Επίσης υπάρχουν οι φήμες ότι η Ρωσία ε, προτίθεται να αποσύρει την υπογραφή της από τον ενεργειακό χάρτη ε, επειδή ε, δεν επιμένει ε, για ένταξη των ΠΟΕ. Αυτές τις φήμες μπορείτε να τις διαψεύσετε ή να τις επιβεβαιώσετε και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρατε ότι θα πρέπει να παίξει ένα στιβαρό ρόλο σε σχέση με τον Ναμπούκο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση του Ναμπούκο. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Σόλτς. Χωρίς μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγήσεις σας και συμφωνώ ότι μέσω της, και πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας χρειαζόμαστε μια ξέχωρη συνθήκη για την ενεργειακή στρατηγική και αντίληψή μας ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει ήδη από το 2006 στο πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Με τον Αμπούκο πιστεύετε ότι θα πετύχουμε ανεξαρτησία αν παραμείνει η διανομή στην Γκάσπρομ και ε, αν η Ρωσία επιχειρήσει όσο περισσότερο, ε, πολύ περισσότερο να επηρεάσει τις ε, χώρες που, το που προωθούν επίσης πώς κρίνεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ε, ένα ε, σοπέκα αερίου από τη Ρωσία. Και τέλος, ε, σε αντίθεση με την εξάρτηση από τη Ρωσία, ε, μήπως υπάρχει η δυνατότητα, το ενδεχόμενο να περάσουμε σε εξάρτηση από την Τουρκία και να θεωρηθεί ότι το πρόγραμμα ε, που ε, έχουμε είναι διακινδυνευμένο. Ο κύριος Στράσερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή, ευχαριστώ και τον κύριο Σάιρους Βόλσκι για την εξαιρετική προκαταρκτική εργασία που έγινε, ούτω ώστε η νέα Κομισιόν και το νέο Κοινοβούλιο να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε στέρεη βάση. Προκειμένου περί, του θέματος αυτού έχουμε ε, μια σύνθετη κατάσταση με προεκτάσεις πέραν της Επιτροπής μας και νομίζω ότι πρέπει να παρατηρήσουμε γι' αυτό το λόγο ότι γενικά πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή επάρκεια, τους ιδίους πόρους μας και θα πρέπει να ε, έχουμε εφοδιασμό πρόσθετο είτε πρόκειται για, τον Αμπούκο ή για άλλους αγωγούς. Και χρειαζόμαστε πολλούς προμηθευτές, ούτω ώστε να μην ε, έχουμε εξάρτηση από έναν. Καθοριστική συμβολή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ε, παίζει εξωτερική πολιτική προφανώς και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο όχι μόνο να μιλάει με μία φωνή η Ευρώπη, όπως είπατε πολύ σωστά και όπως προβλέπετε και στην πολιτική σας, αλλά να είναι σε ισότιμη βάση στις συνομιλίες με τους εταίρους. Θα καταστεί απαραίτητο να προχωρήσουμε ε, προς τη Ρωσία ε, με εταιρικό αλλά πολύ ε, στιβαρό τρόπο και η Ρωσία θέλει πράγματα από την Ευρώπη ε, και θα πρέπει να υπάρξει ένα δούνε και λαβίν. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον Κάφκασο, την Κεντρική Ασία, το Ιράν, το Ιράκ και είναι καλό ότι παίζεται νέο ρόλο και στις μεσογειακές χώρες γιατί και αυτό θα βοηθήσει ε, στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Ευχαριστώ. Πάλι για 1,5 λεπτό ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Σήμερα το πρωί, ενώ εσείς κάνατε την παρουσίασή σας, ο κύριος Πίμπολκ ήταν στην Επιτροπή Ενέργειας. Μπορεί να συμβεί αυτό, δεν το επικρίνω, αλλά καλό είναι να συντονίζομαι καλύτερα τις ε, δραστηριότητες των επιτροπών μας, γιατί αυτό είναι σημαντικό θέμα και για τις δύο επιτροπές και πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή κοινοβουλευτική εξέταση του θέματος. Δεν φταίτε εσείς κύριε Λανταμπούρου ή κάποιος άλλος, αλλά να αποφεύγονται τέτοια πράγματα στο μέλλον. Δεύτερη παρατήρηση, Ναμπούκο και South Stream. σχεδιασμός άνοιγμά του. Θα ήθελα τη γνώμη της Κομισιόν, όχι τώρα κατά ανάγκη, αλλά ίσως στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ε, ίσως οι Κομισιόν είναι ουδέτεροι και δεν θέλουν να δώσουν προτεραιότητα και προτίμηση σε έναν αγωγό. Αλλά θα θέλαμε τουλάχιστον τη θέση της Κομισιόν σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Όπως είπατε, μία ιδέα είναι η μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία. Όχι ότι μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι, ε, ε, το ρωσικό αέριο. Αυτό δεν έχει νόημα, αλλά τουλάχιστον να δοθεί μια προτίμηση στον Αμπούκο. Να δούμε το θέμα των τιμών, ε, τα θέματα της διεύρυνσης. Κάποιες παρατηρήσεις θα, ήταν, θα είναι ουδέτερη, έχει κάποια προτίμηση κομισιών ή έχει κάποια χρονική προτίμηση. Κάποιες λεπτομέρειες θα ήταν ενδιαφέρουσες πάνω σε αυτό το θέμα χωρίς να θέλω κατά ανάγκη να πείτε ότι το ένα είναι καλό και το άλλο κακό. Ευχαριστώ. Ο Βάιγκελ, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως είναι σημαντικό το γεγονός ότι πολλή προσοχή έχει δοθεί στις σχέσεις με τη Ρωσία στα πλαίσια της πολιτικής ενέργειας. Σαφώς αυτό είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για να δούμε την συνολικότερη πολιτική μας με τη Ρωσία. Και βεβαίως πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις βελτιώσεις που απαιτούνται ε, εκεί. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα της έρευνας. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι αυτά δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό της ενεργειακής ασφάλειας. Έχω υπόψη με εδώ το Τουρκμενιστάν, για παράδειγμα, που είναι από τις χειρότερες δικτατορίες στον κόσμο. Και τη Ρωσία μπορούμε να την βάλουμε εδώ, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή. Ποια είναι η δική σας γνώμη, παρακαλώ, στο θέμα αυτό. Πώς μπορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να αντιμετωπιστούν καλύτερα ε, στην εξωτερική πολιτική ενεργειακή ασφάλειας που διαμορφώνεται τώρα ώστε τα θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφάλειας να μην αντιμετωπίζονται ξέχωρα αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα. Και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ενεργειακοί μας εταίροι ε, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας Τώρα ε, θα κατασκευαστεί ο αγωγός Nord Stream. Φαίνεται πολύ δυσχέρης η όλη κατάσταση γιατί είναι σαφές ότι οι χώρες ε, που ενέχονται δεν εμπιστεύονται μία στην άλλη. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Η Ρωσία για παράδειγμα δεν έχει δεσμευτεί σε μια διεθνή συνθήκη που λέγεται η συνθήκη ΕΣΠΟ και αφορά τις... Ε, ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ανάλυση τους όταν πρόκειται για διασυνοριακά έργα. Δεν πρέπει λοιπόν να δεσμευτούν και να υπογράψουν αυτές τις διεθνείς συνθήκες που πρέπει να την χάνουν σεβασμού όταν γίνονται τέτοια προγράμματα. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ο κύριος ε, Σόλτσε από την ε, Νοτική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Γενική Διευθυντά πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, η ενέργεια δεν θα πρέπει να ε, καταναλώνεται άσκοπα ε, και να σπαταλάτε. μιλάμε για FEE e. Ε, χρησιμοποίηση ενέργειας. Τι ρόλο παίζει στι τωρινέ διαπραγματεύσεις αυτή. Επίσης, ε, ενεργειακός εφοδιασμός ε, με βάση σωστέ εταιρικέ σχέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, Ναμπούκο, ο South Stream, ο αγωγό της Βαλτική, το Euromed κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα που πολλές φορές ε, δεν ε, τα προσεγγίζομαι ε, από κοινού. Πώς μπορούμε λοιπόν από κοινού με τις χώρες εταίρους μας να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακό εφοδιασμό σαν άμεση προοπτική στην πολιτική μας. Ευχαριστώ τον κύριο Σόλτς. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, θα ήθελα να ρωτήσω για τη Ρωσία και τον ενεργειακό χάρτη. Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε στην Επιτροπή την, ε, τον ενεργειακό χάρτη και τα πράγματα πάνε, ε, εξελίσσονται αρνητικά. Η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει το χάρτη, ε, πρέπει να επικυρωθεί υποτίθεται στα ψηφίσματα και σε άλλα κείμενα ε, υπογραμμίζεται ότι είναι δεσμευτικός ο χάρτης για τη Ρωσία και υπάρχει και μια ειδική παράγραφος 45 ίσως ε, που αναφέρει ρητά ότι ε, το θέμα αυτό τώρα χρησιμοποιούν οι ρωσικές αρχές ένα άλλο επιχείρημα ότι δηλαδή αναγκάστηκαν ε, να υπογράψουν την εποχή που η Ρωσία ήταν ε, αδύναμη χώρα, τώρα είναι ισχυρή και δεν είναι πια δεσμευτικό. Αυτό λέει πολλά ως παράδειγμα για το μέλλον. Ε, επίσης, με ομό τρόπο είπαν ότι δεν θα την, τον εφαρμόσουν αλλά θα παρουσιάσουμε το δικό μας σχέδιο και θα υπογράψετε εσείς το κείμενό μας. Πρόσφατα, επίσης, απέσυρε την υπογραφή και αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν να επιβάλλουν στην Ευρώπη τους δικούς τους όρους. Εσείς ε, κύριε Γενικέ Διευθυντά ε, το έχετε αυτό το νέο ρωσικό σχέδιο κειμένου που θέλουν να επιβάλλουν στην Ευρώπη ή δεν το πήρατε ακόμη. Ευχαριστώ κύριε Λανσμπέργκης και τώρα ο συνάδελφος ένα 1,5 λεπτό. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά για την ε, ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την Αρκτική, όπου λαμβάνουν χώρα ταχύτατες αλλαγές πιο ταχείες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός ενεργειακός στην αρκτική περιοχή. Η Κομισιόν ακόμη δεν έχει αποφανθεί. Ε, εξετάζει το θέμα. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να βάλουμε ε, στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας στην Αρκτική όταν μιλάμε για θέματα ενέργειας. Επίσης, η ερώτηση της κυρίας ε, Χάουταλα για το North Stream αγωγό. Πολλές περιβαλλοντικές μελέτες έχουν γίνει για το πρόγραμμα αυτό όπως και σε άλλα ενεργειακά προγράμματα. Πιστεύετε ότι στο North Stream θα πρέπει να δούμε θέματα ασφάλειας και όχι μόνο τα περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ. Γιατί που είσαστε τόσο σύντομοι. Και τώρα η κυρία Λούνατσεκ, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λανταμπούρου, πολύ σωστά και αναγκαστικά μας είπατε πόσο θα βοηθήσει η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας αφού αν θέλετε θα υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Απαραίτητο είναι αυτό, το είδαμε και τώρα. Ήδη κάποιοι προλαλήσαντες ανέφεραν τον κατακαιρματισμό της ενεργειακής πολιτικής των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν πράγματι νομίζω ότι θα είναι αναγκαίο και θα βοηθήσει η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας για κοινή στρατηγική σε ενεργειακά θέματα. Τώρα, αν θα έχουμε επιτυχία αυτό θα το δείξει το μέλλον. Εγώ θέλω να κάνω μια ακόμη ερώτηση ε, που ήδη αναφέρθηκε. Ε, είπατε πόσο σημαντικό είναι να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία. Συμμερίζομαι την άποψη αυτή. Εμείς τη συμμεριζόμεθα την άποψη αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια εσείς και η Κομισιόν πώς κρίνετε το γεγονός ότι στην Αυστρία αυτή η ε, ε, η Baumgarten έχει συμμετοχή 50% της Gazprom γιατί ε, αυτή η πλατφόρμα είναι σημαντική αλλά έχει συμμετοχή 50% η Gazprom εκεί. Αυτό είναι προβληματικό. Πάντω είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα της εξάρτησης ε, ή της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία έτσι περιορίζεται. Θα με ενδιαφέρε πώς βλέπει η Κομισιόν το θέμα αυτό και τι θέση ε, παίρνει επί του ζητήματος. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Ο κύριος Κέλλαμ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λανταμπούρου, ευχαριστώ για τα εντυπωσιακά σας επιτεύγματα στον τομέα της ενέργειας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας στο μέλλον. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εμπιστοσύνη στην Κομισιόν μέσα από το έργο της. Είναι σημαντικό αυτό. Συμφωνώ με την αναφορά σας στον Ζακ Ντελόρ χρειάζεται η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και μια ενεργειακή συνθήκη δεσμευτική για μας. Αλλά ε, επειδή στηριχθήκαμε στην ε, έκθεση πριν από δύο χρόνια Cyrus Walls και θα ήθελα να ε, κάνω δύο ερωτήσεις. Η Άφετ θεωρεί ότι η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει μέτρα ούτως ώστε να περιορίσει ανεξέλεγκτες επενδύσεις κρατικών εταιριών ε, στον ενεργειακό τομέα. Στο μέλλον, ε, εμπορικές συμφωνίες με τρίτους εταίρους ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και ρήτρες ενεργειακής ασφάλειας. Αυτές οι προτάσεις ευδοκίμησαν και σε ποιο βαθμό. Τι μπορείτε να μας πείτε τώρα που θα φύγετε από την Κομισιόν. Επίσης, συμφωνώ με τη συνάδελφο Χάουταλα ε, ότι στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον Nord Stream θα πρέπει να επιβάλλουμε τον όρο να ε, δεχτεί την ε, σύμβαση ΕΣΠΟ η Ρωσία. Κύριος Κασουλίδης, παρακαλώ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για κοινή ενεργειακή πολιτική ε, ανοίγονται ρεαλιστικές προοπτικές. Ε, ε, η κοινή ενεργειακή πολιτική διαφοροποιείται γιατί υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες στο ενεργειακό μίξ κάθε χώρας. Δύο ερωτήσεις. Πόσο ρεαλιστικό είναι να έχουμε ενεργειακή συμφωνία με την Ρωσία πάνω στην αρχή της του ασφαλούς εφοδιασμού ε, ενέργειας και της ε, ε, προσφοράς ζήτησης. Δεύτερον, πόσο έχουν προχωρήσει τα σχέδιά μας που λαμβάνουν υπόψη το θέμα της αλληλεγγύης, αν υπάρχει ενεργειακή κρίση, ενεργειακή διαφοροποίηση, τα διαφορετικά υφιστάμενα δίκτυα, ούτω ώστε να υποστηριχθεί μια χώρα που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, και το θέμα ε, της ε, αποθήκευσης ε, LNG υγρού αερίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάντεμπουρου έχει το λόγο για να απαντήσει στη σωρία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε ως προς αυτό το θέμα και για τις ε, ιδιαίτερα οξυδερκείς ερωτήσεις που υποβάλλατε. Σε αυτό το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, ε, δεν ε, έχω την αξίωση να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις λεπτομερώς. Θα προβώ σε ορισμένα σχόλια ως προς τα θέματα που εθίγησαν, δηλαδή τα βασικά θέματα βάσει των ερωτήσεων και εάν δεν έχω απαντήσει συγκεκριμένα στα, στο ερώτημά σας, θα ήθελα να μου την υποβάλλετε γραπτός και με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε ερωτήσεις μία προς μία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπεκφεύγω των ευθυνών μου και θα σας απαντήσω συγκεκριμένα σε όλες τις ερωτήσεις αν μου στείλετε ένα email. Ποια είναι τα θέματα που διέπουν τις ε, ερωτήσεις σας. Σε πολλές από τις ερωτήσεις ανακύπτει το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία. Πρώτο σχόλιο. Καθίσταται σαφές ότι οι σχέσεις μας με αυτή τη χώρα στον τομέα ενεργειακής συνεργασίας πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής έναντι αυτής της χώρας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η χώρα αυτή είναι μια ε, γείτον χώρα, δεν, έχουμε πάντα, δεν είχαμε πάντα τις καλύτερες ε, δυνατές σχέσεις, τις καλύτερες, ε, δεν τις αναπτύξαμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά εδώ και ένα χρόνο στην αξιολόγηση και στην ιεράρχησή μας θεωρήσαμε ότι η αλληλεξάρτηση είναι τέτοια, τα γεωπολιτικά μας ε, συμφέροντα είναι τέτοια που θα πρέπει να εξεύρουμε ε, τρόπους διαλόγου και συνεργασίας. Ακόμα και εάν δεν μας είναι ε, οι συμπαθείς ή οι θύνοντες αυτής της χώρας. Το θέμα της ενέργειας είναι πρώτη τη σημασία. Χρειαζόμαστε τη Ρωσία, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική βραχυπρόθεσμα στην προμήθεια φυσικού αερίου. Χρειαζόμαστε μεγάλες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ούτε η Νορβηγία ούτε η Αλγερία δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία δεν μας χρειάζεται. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα μπορούσε να ε, πωλήσει τα προϊόντα της φυσικού αερίου και πετρελαίου σε μια τόσο μεγάλη οντότητα όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σε τελευταία ανάλυση μπορεί να λέγεται ότι δεν μας χρειάζεται, αλλά επί της ουσίας μας χρειάζεται. Αυτή η αλληλεξάρτηση είναι υπαρκτή, γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας, θα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι, να μιλάμε με μία φωνή και επειδή είμαστε δυνατοί θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις θέσεις και τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους Ρώσους εάν δεν λάβουμε υπόψη τις δικές μας θεμελιώδεις αξίες. Και όπως είπατε κυρία μου και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει για τη Ρωσία αλλά και για όλες τις χώρες. Και για να έχουμε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία αναχείρας για να προωθήσουμε μια ε, συνεπή στρατηγική. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, διότι θα πρέπει οι πολίτες μας να έχουν την δυνατότητα να παραγούν, ε, να έχουν επαρκή θέρμανση, να μπορέσουν να πολεμήσουν, να καταπολεμήσουν τους εξωγενείς κλιματικούς παράγοντες, αλλά αυτό μέσα στα πλαίσια των αξιών μας. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κοινοβούλιο, αυτό πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση και ένα θεσμικό όργανο όπως η Εκτελεστική Επιτροπή, διότι η πραγματικότητα αυτή είναι. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε υποχωρήσεις, είτε στον ένα τομέα ή στον άλλο. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη ασκούν μεγάλη πίεση για μία συμφωνία σύνδεσης με την Αρμενία, Γεωργία και Αζερβαϊτζάν για τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου. Μέχρι τώρα είπαμε ότι δεν θα ξεκινήσουμε καμία διαπραγμάτευση εάν σε μια συγκεκριμένη χώρα, στο Αζερβαϊτζάν, δεν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης ως προς την ε, λειτουργία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουμε με το Συμβούλιο και θα πρέπει να εξεύρουμε μια ισορροπημένη λύση. Επειδή ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, γνωρίζω ότι υπάρχει αξιοπιστία στην Ευρώπη, ως προς την Ευρώπη, διότι επιβάλλει αρχές όπως την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Υπάρχει μεγάλη ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων προς την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν είναι εύκολο είναι να προωθήσουμε μία συνεπή πολιτική προωθώντας τα οικονομικά και εμπορικά μας συμφέροντα σε, ε, σχέση με τα ανθρώπινα, σε συσχετισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως δεν υπάρχει πάντα ε, λύση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με μικρά βήματα όπως πάντα. Επανερχόμενο στη Ρωσία. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία για ένα πλαίσιο συνεργασίας, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Αυτή είναι μια ερώτηση που μου Σε λίγους μήνες. σε, μάλλον για να το θέσω πιο ρεαλιστικά, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Διότι θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις, ε, όχι στα πλαίσια έντασης. Εάν μπορέσουμε στους επόμενους μήνες να φτάσουμε σε μια βελτιωμένη συνεργασία με αυτή τη χώρα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ. Τι αναζητά αυτή η χώρα σε σχέση με εμάς. αναζητά μια συμφωνία ασφαλείας. Ο κύριος Μέτβετεφ το έθεσε αυτό ένα χρόνο πριν στο ΕΒΙΑΜ. Αυτό είναι και μια ιδεολειψία, μια αιμονή και ανάλογα με την απάντησή μας μέσα στα πλαίσια μιας γενικής συμφωνίας ασφάλειας, θα δούμε κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα και μεγαλύτερη ευελιξία για να φτάσουμε σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Για να το πούμε με λίγα και απλά λόγια. Η ενεργειακή συμφωνία με τη Ρωσία δεν εξαρτάται από ενεργειακά ζητήματα και μόνο. Εξαρτάται από μεγαλύτερα και διευρυμένα συμφραζόμενα, πολιτικά συμφραζόμενα. Γι' αυτό αν αφήσουμε κατά μέρος όλες τις εντάσεις με αυτή τη χώρα, και είναι πολλές και μεγάλες, και τις δυσκολίες που έχουμε με αυτή τη χώρα που είναι ε, μεγάλες και πολλές, τεχνικά υπάρχει ε, αμοιβαίο ενδιαφέρον να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Η Ρωσία τι επιθυμεί, τι αναζητά. Θα ήθελε οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν, να αγοράσουν ε, μία συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου και πετρελαίου έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις στη Ρωσία για τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού δικτύου. Δηλαδή, αν δεν έχουν τα χρήματα από την Ευρώπη, τότε οδηγούνται στο χάος. Εμείς, μέσω πρόθεσμα, θέλουμε μία ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή ε, την παροχή συγκεκριμένων ποσοτήτων με συγκεκριμένη τιμή αντίτιμο. Εάν διευθετηθεί αυτό το θέμα, εκείνοι χρειάζονται επενδύσεις για να εξυγχρονιστούν και εμείς χρειαζόμαστε ενεργειακή προμήθεια. Αλλά η ζωή είναι ακόμα είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Προσωπικά και από την πείρα μου ε, θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο και είμαι αισιόδοξο διότι υπάρχει Ε, μία ε, ρεάλ πολιτικ που προωθεί η ρωσική ε, νομενκλατούρα, αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, και αυτό αφορά και τον Πούτιν που θέλει να προβάλλει την εικόνα μιας ισχυρής Ρωσίας, αλλά υπάρχουν και πολιτικοί που θέλουν να εξυγχρονίσουν τη χώρα και θέλουν να εξυγχρονίσουν και τη, χώρα ε, μέσω ενός ανοίγματο. Και τώρα επανέρχομαι στο θέμα του ενεργειακού χάρτη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή μιλήσαν οι Ρώσοι για ένα συμβασμό, τώρα δεν θέλουν όμως να ακυρώσουν την ενεργειακή χάρτα. Τώρα όμως που έχουν αυτή την ενεργειακή δύναμη θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους συλλογιστική. Δεν θα το δεχτούμε εμείς αυτό, διότι εμείς ε, θα διαδραματίσουμε το ρόλο μας γιατί οι Ρώσοι θέλουν να επιβάλλουν στις χώρες διαμετακόμισης όπως την Ουκρανία ε, όρους ελέγχου που δεν ε, περιλαμβάνονται στη χάρτα και θέλουν να μετονομάσουν ορισμένες χώρες ως χώρες διαμετακόμνησης. Δηλαδή, ο κύριος Πούτιν εδώ και πολλά χρόνια θέλει να δημιουργήσει συνθήκες εξάρτησης της Ευρώπης ως προς την αγορά φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δηλαδή, να μας υπεξαιρέσει κάθε δυνατότητα εναλλακτικής λύσης για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή εξάρτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την στρατηγική ελέγχου από πλευράς Ρωσίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μέσω του ανοίγματο νέων δυνατοτήτων προμηθειών. Με το South Stream με τις ε, χώρες που θα μπουν στον Ναμπούκο. Η Ρωσία, κάποιος το είπε εδώ, η Γκάσπρομ βρίσκεται στην κοινοπραξία του Ναμπούκο. Αυτό όμως δεν είναι το πιο βασικό. Το Τουρκμενιστάν, το Αζερβαϊτζάν και το Ουσμπεκιστάν μπορούν να μας προμηθεύσουν τις ενεργειακές ποσότητες για να μειώσουμε την ένταση και την εξάρτηση από τη Ρωσία. Υπάρχουν τρία προβλήματα με τον Αμπόκο. Το πρώτο είναι η δέσμευση αυτών των χωρών της Κεντρικής Ασίας και του Νοτιού Καυκάσου να δεσμευτούν ως προς ενεργειακές ποσότητες που θα μπορούσαν να απολύσουν προς την Ευρώπη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι τώρα. Για με το Αζερβαϊτζάν ισχύει, με το Τουρκμενιστάν όχι, γιατί το Τουρκμενιστάν έχει μεγάλες δυσχέρειες με τη Ρωσία ως προς εξωτερικές σχέσεις. Το Τουρκμενιστάν βεβαίως δεν είναι δημοκρατική χώρα, αλλά θα ήθελε και προβάλλει μια στρατηγική ενεργειακής ε, διακλάδωσης και διαφοροποίησης. Το ίδιο ισχύει με το Ουσβεκιστάν. Έτσι θα πρέπει να προσδώσουμε αξιοπιστία στο Ναμπούκο. Εμείς θα πρέπει να δεσμευτούμε να αγοράσουμε συγκεκριμένες ποσότητες. Δηλαδή, για ποιες ποσότητες ε, δεσμευόμαστε ως προς αυτές τις χώρες. Η κατάσταση βελτιώνεται. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα της διαμετακόμισης. Και επανέρχομαι με το θέμα του ότι στις 8 Μαΐου στην Πράγα έγινε μία διάσκεψη με όλες αυτές τις χώρες όπου είχαμε μία απαρχή δέσμευσης ως προς αυτά τα θέματα που θα πρέπει να επιληθούν για να καταστεί αξιόπιστο το Ναπουκό. Μετά είχαμε μία διακυβερνητική ε, συμφωνία όπου οι Τούρκοι δεσμεύτηκαν για πρώτη φορά να θέσουν σε εφαρμογή διαμετακομιστικούς μηχανισμούς που να είναι καλοί και για μας και για τους προμηθευτές. Δηλαδή, δεν θα ε, προσλάβουν ένα μέρος του φυσικού αερίου για ίδια κατανάλωση και ε, διαμέσου αυτής της διαμετακόμισης από τη χώρα τους θα, μπορέσουν, θα λάβουν μια ποσότητα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. Ήταν πολύ σημαντική η δέσμευση των Τούρκων τον Ιούλιο, διότι έτσι το Ναμπούκο καθίσταται πιο αξιόπιστο άλλη καινοτομία του Ναμπούκο. Το Ιράκ δεσμεύτηκε για προμήθεια ποσοτήτων στην Ευρώπη μέσω του Ναμπούκο. Άρα, σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη από εδώ και τρεις μήνες. Χρειάζονται ευρωπαϊκά κονδύλια, πιστώσεις. Αυτό εξαρτάται από εσά, κυρίες και κύριοι. Εσείς είσαστε ένα σκέλος της δημοσιονομικής αρχής. Εάν στη δημοσιονομική συζήτηση θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει, θα το κάνει. Και στον παρόντα προϋπολογισμό υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν επαρκούν για να προωθηθεί το Ναμπούκο. Άρα το θέμα του Ναμπούκο είναι ανοιχτό, έχει υψηλότερη αξιοπιστία σε σχέση με τρεις μήνες πριν ή μερικά χρόνια πριν. Τώρα, σχέσεις South Stream και Ναμπούκο. Εμείς, κύριε Σπόποντα ήταν δική σας η ερώτηση. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολλαπλασιασμός πηγών ενεργείας και προμήθειας είναι καλός. Δεν είμαστε κατά του South Stream, ούτε το θέτουμε σε ανταγωνιστικές σχέσεις με τον Ναμπούκο. Εγώ λέω, σας λέω ειλικρινά, προτιμώ το Ναμπούκο, διότι μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, κατά το οποίο δεν κάνει ο άλλος διάδρομος. Και η Ιταλία πριν να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνίες με τη Ρωσία, σε σχέση με αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα θα έπρεπε να μας είχε συμβουλευτεί. Κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζουμε καμία συμφωνία, καμία σύμβαση των κρατών μελών σε σχέση με αυτό το δίκτυο προμηθειών. Γνωρίζουμε το deal, το έγγραφο που υπάρχει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Καμία χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ζητήσουμε από τη Γαλλία, από την ε, Ιταλία και από την Γερμανία να μας δώσουν ε, αντίγραφα της συμφωνίας, δεν το κάνουν. Αυτό δεν το κάνω για να εκφράσω απλώς το παράπονό μου, αλλά για να πω ότι έχουμε να διανύσουμε πολύ μακρύ δρόμο για να έχουμε την ε, δυνατότητα να προωθήσουμε αυτά τα σχέδια ο καθένας κρατά τις πληροφορίες του, διότι υπάρχει αυτή η νοτροπία από αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική. Όλες οι χώρες σκέφτονται τα εθνικά τους συμφέροντα. Και στην ουσία δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δέσμευση. Γι' αυτό πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο. Και συμφωνώ με τον κύριο Σάριους Βόλσκι όταν λέει ότι πολλά έχουν γίνει εξαιτίας και της έκθεσής του, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για τις ε, κατάλληλες, τις σωστές υποχωρήσεις από αυτά. Παραμένω εδώ κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε αυτό τον διάλογο και στο μέλλον, διότι τα θέματα είναι πολλά. Έχουμε να κάνουμε με μια πολυσχηδή πραγματικότητα και θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες δεσμεύσεις στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαντεμπούρου για την αναλυτική του προσέγγιση και παρουσίαση και για τις τελικές απαντήσεις Ξεκινήσαμε με μια καθυστέρηση 20 λεπτών και έχουμε μια πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα εξ ονόματος όλων να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε αυτά τα χρόνια και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και για τη διεύρυνση. Έχετε μια πολιτική με όραμα. Νομίζω ότι ήσασταν βασικός πρωταγωνιστής στην ευρωπαϊκή σκηνή και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο αυτό τρόπο στη νέα σας θέση. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Μαρόκο. Όπως είδα, είπα ήδη στην αρχή της συνεδρίασης, ένα έγγραφο έχει διανεμηθεί. Πρόκειται για ένα σχέδιο ε, προφορικής ερώτησης για την ενεργειακή πολιτική. Εν τω μεταξύ, ενώ είχαμε τη συνεδρίασή μας, υπήρξαν διάφορα αιτήματα τα οποία εκφράστηκαν από μέλη της Επιτροπής ούτω ώστε να τροποποιήσουμε κάπως αυτήν το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Θα σας μόλις θα σας το δώσουμε και πάλι ε, στην συνάντηση των συντονιστών. Τώρα περνάμε ε, στο επόμενο θέμα. Έχουμε τον κύριο Μαρινέσκο που ήταν επικεφαλής ε, της Αντιπροσωπείας Παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές στη Μολδόβα που έλαβαν χώρα μεταξύ 26ης και 30ης Ιουλίου 2009. Και ως προς το θέμα της Μολδαβίας η Επιτροπή μας σε τρεις ευκαιρίες συζήτησε το θέμα μετά από τα γεγονότα των βουλευτικών εκλογών της 5ης Απριλίου. Το θέμα αυτό ε, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε ότι στις 30 Ιουλίου η Διεθνής Αποστολή Παρατηρητών, όπου συμμετείχε και η η δική μας αντιπροσωπεία υπό τον κύριο Μαρινέσου, που διοργάνωσε ο ΑΣΕ, παρακολούθησε αυτή την εκλογική διαδικασία αλλά ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις για την δυνατότητα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε αυτές τις διαδικασίες. Σας παρακαλώ, αν έχετε σχόλια μεταξύ σας, να τα κάνετε εκτός αίθουσας, έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να παρακολουθήσει τις συζητήσεις εντός. Λοιπόν, Δίνω το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αντιπροσωπεία παρατηρητών. Θα μας πει για τις καταγγελίες που έγιναν στη Μολδαβία σε σχέση με, τις, με τη διενέργεια των εκλογών και θα θέλαμε ένα γενικότερο σχολιασμό ως προς την, ε, τις πολιτικές εξελίξεις στη Μολδαβία, ιδιαίτερα ως προς σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, στις 29 Ιουλίου είχαμε εκλογές στην Δημοκρατία ε, της Μολδόβας λόγω ε, της αποτυχίας του Κοινοβουλίου να εκλέξει ένα νέο πρόεδρο μετά τις εκλογές, διότι αυτό προβλέπει το Σύνταγμα ε, της Μολδόβας, δηλαδή μια επανάληψη των εκλογών. Όπως ξέρετε, έχει ε, γίνει δεκτή η δημιουργία μιας ε, ομάδας παρατηρητών. Είχαμε 7, 3 από το ΕΛΚ, εγώ ίδιος, ο κύριος Τσίπ, ο κύριος Μπρέντα, δύο εκπρόσωποι από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κ. Μπαλτσίτης από τη Λιθουανία και ε, κάποιος από την Βουλγαρία, ένας εκπρόσωπος ε, της ε, Άλντε της Ρουμανίας και εκπρόσωπος των Πρασίνων από τη Λετωνία. Στις 27 και 28 Ιουλίου συναντήσαμε τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδόβα, τον κύριο Τσέσαρε Ντιμόντι και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων στη Μολδόβα και τον ε, ύπατο εκπρόσωπο ε, Κλάτμαν Μίτσεκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδόβα. Λάβαμε μέρος σε όλες τις αποστολές που οργανώθηκαν από την Διεθνή Ομάδα Παρατηρητών. Συναντήσαμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, μέσα ενημέρωση, στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ε, βασιστήκαμε σε προκαταρκτικές εκθέσεις ε, παρατηρητών και μπορέσαμε να εξαγάγουμε τα κόλτα συμπεράσματα σε σχέση με τις εκλογές που έλαβαν χώρα την 5η Απριλίου. Το ε, κατόφλι μειώθηκε από 6 σε 5% το εκλογικό μέτρο και η ανάγκη 50% συμμετοχής μειώθηκε σε 35%. Ωστόσο, περιορισμοί ως προς τα εκλογικά δικαιώματα διατηρήθηκαν ε, και επίσης ε, διατηρήθηκε ο περιορισμός ως προς τα άτομα που είχαν πολλαπλή ηθαγένεια. Είχαμε αμοιβέ ε, επιθέσεις ε, μεταξύ των κομμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ήταν πίσω από, την εξε... από τις ταραχές και το ίδιο και η, αντιπολίτευση για τους κομμουνιστές. Υπήρχε επιθετικότητα ακόμα και εχθρότητα που οδήγησε σε πόλωση της κατάστασης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποίησε τις διοικητικούς πόρους της κυβέρνησης για να ασκήσει πίεση και να εκφοβήσει κυρίως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση, κυρίως τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, είχε δυσανάλογη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατάφεραν να έχουν κάποια πρόσβαση στα μέσα πράγμα που δεν είχε γίνει στις εκλογές της 5ης Απριλίου. Ε, σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους, ε, κανένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν τον Απρίλιο ε, δεν επιλύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι κατάλογοι και η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να ενημερωθούν οι κατάλογοι. Μόνο 33 εκλογικά τμήματα οργανώθηκαν έξω που είναι ανεπαρκέσλο υπάρχει μεγάλος αριθμός υπηκών της Μολδόβας που ζουν στο εξωτερικό, μεταξύ 600.000 έως και 1 εκατομμύριο σύμφωνα με τις πληροφορίες Μαριαν Λούκου, πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτομόλυσε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και ίδρυσε ένα δημοκρατικό κόμμα με το οποίο παρουσιάστηκε και πέρασε το μέτρο το εκλογικό, το κατόφλι ε, Είχαμε τέσσερις ομάδες ε, και πήγαμε σε 40 έως 50 εκλογικά τμήματα. Δεν σημειώσαμε μεγάλες παρατυπίες εκτός από προβλήματα με τους εκλογικούς καταλόγους, άτομα ε, που βρισκόντουσαν στους καταλάγους και δεν θα έπρεπε να είναι. Ε, κοινοποιήσαμε αυτές τις παρατυπίες στις αρχές σχετικά με τα προβλήματα αυτά οι ε, υπηκόοι της Μολδόβας που ζουν στην υπερδνηστερία μπορούσαν να ψηφίσουν ε, στην δυτική όχθη του Δνίστερου ε, και πάρα πολύ λίγοι από αυτούς επέλεξαν αυτή τη λύση. Τα αποτελέσματα ήταν Κομμουνιστικό Κόμμα, 48 έδρες στο Κοινοβούλιο, 12 ε, λιγότερες από τον Απρίλιο, Δημοκρατικό Κόμμα 18, αύξηση κατά τρία ε, σέντρες, η φιλελεύθερη 15, τη ίδια ποσότητα, Δημοκρατικό Κόμμα 13 και Μολδόβα Νάστρα Συμμαχία 7 έδρες στο Κοινοβούλιο, 5 λιγότερες από ό,τι τον Απρίλιο. Μερικές σύντομες ε, παρατηρήσεις και ε, συμπεράσματα νομοθετικές αλλαγές πρέπει να γίνουν για πιο δίκαιες εκλογές στο μέλλον. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να υπάρχει ο κατάλογος των πολιτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Ούτως πρέπει να υπάρχει και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα ε, το το φιλελεύθερο κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και η Συμμαχία Μολδοβανόστρα έχουν δημιουργήσει έναν συναπισμό που είναι ε, ο συνασπισμός, η Συμμαχία για την Μολδόβα και τον Αύγουστο εξέλεξαν έναν πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μιχαήλ Γκίμπου, που είναι ο πρόεδρος της φιλελεύθερου, φιλελεύθερου κόμματος. Σήμερα θα προσπαθήσουν να εκλέξουν ένα νέο πρόεδρο της χώρας, αλλά Αυτές οι 53 έδρες που έχουν στο Κοινοβούλιο δεν υπαρκούν για να εκλέξουν τον πρόεδρο της Μολδόβας. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 61 ψήφους. Ο υποψήφιος για πρωθυπουργό είναι επικεφαλής του Δημοκρατικού και ο κύριος Μαριάν Λούπου θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Εάν αποτύχουν να έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 ψήφων, θα πρέπει να οργανώσουν νέες εκλογές το 2010. Ό,τι και να συμβεί, η δημοκρατία της Μολδόβας θα χρειαστεί ε, μεγάλη υποστήριξη ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις ε, που την ταλανίζουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί για να στηρίξει την δημοκρατία της Μολδόβας τους επόμενους μήνες ε, ε, καταληκτικά θα ήθελα να πω ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ενταχθεί στην ε, Διεθνή Αποστολή Παρατηρητών με την αντιπροσωπεία του ΑΣΕ και του ΙΣΥ. Όταν αρχίσαμε τη συζήτηση για την προκαταρκτική έκθεση ο κύριος Πέτερς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ, κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έλλειψη ε, πίστης ε, και εξέφρασε ε, μία δυσπιστία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή ε, είχαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στη Μολδόβα του Μαΐου 2009 και κυρίως το άρθρο 22 το οποίο και Παραθέτω λέει ότι οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην έκθεση την προεκτατική του ΟΑΣΕ σύμφωνα με τις, για εκλογές του Απριλίου και, ή τους, ε, και ισχυρισμούς πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων σχετικά με τις υποτιθέμενες παρατυπίες σε αυτές τις εκλογές και τονίζει ότι αυτές οι διαφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ΟΑΣΕ στις μελλοντικές εκλογές και εκθέσεις Τέλος της παράθεσης. Μου λέχθηκε ότι η αντιπρόσωπεία του ΕΛΚΑ θα έπρεπε να συντάξει μια χωριστή έκθεση σχετικά με τις εκλογές με την υποστήριξη του επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορέσαμε ε, να διευθετήσουμε αυτή την αντιπαράθεση. Κάναμε μια ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης και χρειαζόμαστε ε, μια επισκόπηση σχετικά με το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται με άλλα όργανα στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος σε αυτή την αντιπροσωπεία και που συμμετείχαν θετικά στη δραστηριότητα που είχαμε στην δημοκρατία της και ελπίζω ότι θα μου θέσετε ερωτήσει Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων κύριε Μαρινέσκου για την ε, σαφή και πλήρη παρουσίασή σας. Τώρα έχω τέσσερα άτομα που ζήτησαν το λόγο ε, και θα πρέπει να περιοριστούν στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να τελειώσουμε εγκαίρας, γιατί ε, θα μας έρθει στις 11 ο κύριος Όλι Ρεν. Θα κλείσω λοιπόν τη συζήτηση με τους πέντε ομιλητές που έχουμε στον κατάλογο και θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να περιοριστούν σε 1,5 λεπτό, όχι περισσότερο, κύριε Σέντρα. Δεν πρόκειται να μιλήσω για την έκθεση ή για την κατάσταση την εκλογική. Νομίζω ότι είχαμε μια πλήρη παρουσίαση, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για μας, για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο και να υποστηρίξουμε τις θετικές εξελίξεις στη δημοκρατία της Μολδόβας. Νομίζω ότι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους είναι για αυτούς που έχασαν τις τελευταίες εκλογές και που βρίσκονται τώρα που σκέφτονται ότι η αντιπαράθεση είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουν την πλειοψηφία που θα τους επιτρέψει να εκλέξουν τον πρόεδρο και τους άλλους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα υπάρξει μια επιτυχία, αλλά η συνέχιση αυτής της διαδικασίας των πρόωρων εκλογών θα μπορούσε να δημιουργήσει ή και να ενισχύσει την πολιτική αστάθεια στη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι από πολιτικής απόψεως δεν πρέπει εμείς να λάβουμε θέση τώρα, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους όσοι θέλουν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα στη χώρα και να αφήσουμε κατά μέρο όσους στο παρελθόν δεν εργάστηκαν για την εδραίωση της δημοκρατία στην Μολδόβα. Θα πρέπει εμεί να έχουμε ένα πακέτο στήριξη οικονομική για τη χώρα, το οποίο θα επιτρέψει στη χώρα να αποφύγει την κοινωνική αναταραχή που είναι μια μεγάλη απειλή και κίνδυνος. Ε, κλείνω, θα πρέπει να ρωτή, ζητήσουμε από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μας να δραστηριοποιηθούν και να δεσμευθούν περισσότερο ούτως ώστε να δοθεί η τεχνική, η πολιτική βοήθεια και για να προτείνουμε μια, ένα οικονομικό και χρηματοοικονομικό παλέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Λάνσδορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Διάβασα την έκθεση των διεθνών παρατηρητών των εκλογών και λέει πρώτα-πρώτα ότι ε, χαρακτηριστικό εδώ ήταν η αδυναμία του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας να βγάλει πρόεδρο μετά τις εκλογές του Απριλίου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πάλι δείχνει ότι η συνταγματική πλειοψηφία δεν αναμένεται για την εκλογή πρόεδρου και εκπλήσωμε λίγο από αυτό που είπε ο κύριος Σεβερίν που βλέπει θετική εξέλιξη και σταθεροποίηση. Ρωτώ λοιπόν τον παρατηρητή μας πώς εκτιμά την κατάσταση είναι θετική πολιτική εξέλιξη ή έχουμε παράταση της στασιμότητας στην πολιτική αφού δεν γίνεται σχηματισμός κυβέρνησης με τρόπο συνταγματικό. Δεύτερον, μετά τις εκλογές του Απριλίου έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τη διάσταση των σχέσεων Μολδαβίας-Ρουμανίας. Ο τότε πρόεδρος ε, ε, Βορώνινε έδιωξε τον ε, πρεσβευτή, τον απέλασε και ε, ε, φρόντισε να απλουστευθεί η διαδικασία ε, απόκτησης της ρουμανικής ηθαγένειας. τι εξέλιξη δόθηκε στην κατάσταση αυτή. Ε, μας είπατε για τις πολλαπλές ηθαγένειες και ότι τα πράγματα δεν είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Στην έκθεσή σας αυτό όμως είναι ένα από τα σημεία που επικρίνονται γιατί ακόμη δεν έχει ακόμη επαρκώς νομικός ρυθμιστεί το θέμα τι, ε, αποτε... τι, επίπτωση είχε σε αυτές τις εκλογές αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Βιγγέιν. Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα ήμουν μέρος της αντιπροσωπείας παρατηρητών. Θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Σύμφωνα με τις περισσότερες παρατηρητές και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών πολιτικών κομμάτων, οι εκλογές ήταν καλύτερα οργανωμένες από αυτές του Απριλίου, ε, τόσο προεκλογικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών. Και μπορούμε να πούμε ότι κατά το μάλλον ήτον η Μολδόβα το πέρα, της πέρασε αυτές τις εξετάσεις, αυτή τη δοκιμασία. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ότι η εκλογική εκστρατεία δεν βασιζόταν τόσο σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα, αλλά πολύ περισσότερο πάνω στα θέματα που έχουν σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του Απριλίου. Μου φαίνεται ότι ακόμα και τώρα τα πολιτικά κόμματα δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη είναι η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση στην Μολδόβα και η οποία επιδεινώνεται και ταχύτατα. Ρόλος μας θα ήταν λοιπόν να τους ενθαρρύνουμε να βρουν ένα συμβιβασμό. Όπως είπε ο κ. Σέβριν, δεν πρέπει να λάβουμε θέση υπό τον ή τον δε, αλλά να κάνουμε ε, την Μολδόβα να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα της και να την βοηθήσουμε να έχει υπεύθυνα πολιτικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι η Συμμαχία για την ε, Ευρωπαϊκή Ένταξη έκανε βήματα πρόοδου και πρότεινε τον κύριο Λούπου ε, για πρόοδο ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τύχει της υποστήριξης του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά έχουμε και την σημερινή αντιπολίτευση και δεν θα ήταν έκπληξη αν θα έχουμε νέες εκλογές το Φεβρουάριο. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε την απαιτούμενη πίεση ούτω ώστε όλες αυτές οι δυσκολίες στον νόμο και στην προετοιμασία των εκλογών να αντιμετωπιστούν αμέσως, ούτω ώστε αν υπάρξουν νέες εκλογές του χρόνου να μην ξαναεμφανιστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Βιγγένεν. Ο κύριος Βέμπερ έχει τον λόγο. Δύο λεπτά, όχι περισσότερο. Θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομη, συμμερίζομαι ε, τις απόψεις που παρουσίασε εδώ ο κύριος Μαρινέσκου και είναι αληθές ότι όλη η προεκλογική εκστρατεία είχε μεγάλη ένταση, ε, και πολλές άνισες δυνατότητες για τα κόμματα να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούν ακόμη ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει νοθεία, αλλά Υπάρχουν δυνατότητες νοθείας λόγω των εκλογικών καταλόγων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι προσωπικά σε διάφορα μέρη ε, συνήντησα ε, Μολδαβούς ε, οι οποίοι ειλικρινά πιστεύουν ότι χρησιμεύσε η ψήφος τους και νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να συγχαρούμε τον λαό της Μολδόβας για τα αποτελέσματα των εκλογών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναντήσεις που είχαμε και το πώς όλα οργανώθηκαν, θα πρέπει να πω ότι υποστηρίζω την ιδέα ότι στο μέλλον θα πρέπει να δράσουμε διαφορετικά και ε, θα αγωνιστώ για αυτήν την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ε, την δική της αποστολή παρατηρητών ακόμα και στα εδάφη που καλύπτει ο ΑΣΕ. Αν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε ένας σημαντικός πρωταγωνιστής, θα πρέπει να δράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι σε αυτές τις αποστολές και να ακολουθούμε τη δική μας μεθοδολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Και τώρα να κλείσουμε ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Μαρινέσκου. Νομίζω ότι το έργο σας συνέβαλε στη σωστή διεξαγωγή των εκλογών με λίγες ενστάσεις, αλλά είναι προβληματικό το αποτέλεσμα ότι υπάρχει μια κατάσταση στασιμότητας και δεν μπορεί ε, να αλλάξει η κατάσταση. Ε, είναι περίπλοκα τα πράγματα και προβληματικά. Μέχρι τώρα είχαμε 800.000 Μολδαβούς που είχαν τη ρουμανική ηθαγένεια και φαίνεται ότι με την απογοήτευση αυτή η τάση αυξάνεται και σιγά σιγά ε, περνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσω της ρουμανικής ηθαγένειας. Ε, αυτό πώς κρίνεται ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον κύριο Σούλτσο. Και έληξαν οι ερωτήσει Θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, τον δόκτωρα Μπρέντα. Ε, ένα λεπτό παρουσίαση του τι προετοιμάζουμε για να υποστηρίξουμε τη Μολδόβα Έχουμε σημειώσει προσεκτικά τα όσα είπατε και έχουμε πλήρη συνείδηση της σημασίας να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ετοιμάσει ένα πακέτο βοήθειας για τη δημοκρατία, 4 εκατομμύρια ευρώ για μερικές από τα βασικά θέματα, τα οποία τονίστηκαν επίσης στη σημερινή παρουσίαση. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι το πακέτο αυτό ε, θα προωθηθεί σύντομα και θα καλύψει ε, μερικά από τα σημερινά ε, θέματα, η μεταρρύθμιση των μέσων ενημέρωσης, υποστήριξη στον συνήγορο του πολίτη της χώρας και επίσης σε άλλους τομείς που ενέχουν μεγάλη σημασία στα πλαίσια των προσπαθειών μας να βοηθήσουμε τη δημοκρατική μεταρρύθμιση στη Μολδόβα. Δεύτερον, είμαστε Έχουμε πλήρη συνείδηση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και θα δώσουμε μια μακροοικονομική βοήθεια στην Μολδόβα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε ακόμα το ακριβές ποσό, το κονδύλιο για την ώρα για να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά ασχολούμεθα ενεργά με το θέμα και προτιθέμεθα να επανέλθουμε με το θέμα αυτό, με το ακριβές ποσό και θα ήθελα να πω ότι είμαστε έτοιμοι ε, να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης, διότι όπως λέχθηκε στην αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση μας να την εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις όταν θα πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως ο συνάδελφος Μαρινέσκου θα ήθελε να απαντήσει σε ορισμένε παρατηρήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με ε, τις παρατηρήσεις του κυρίου Σούλτς που είπε ότι 800.000 υπήκοοι της Μολδόβας απέτυχαν ρουμανική υπηκότητα. Αυτό είναι ο αριθμός που έχετε. Όχι, δεν είναι αληθινός αυτός ο αριθμός. Είναι περίπου 30-40.000 ε, ε, ηθαγενείς της Μολδόβας που πήραν την ρουμανική υπηκότητα τα 20 τελευταία χρόνια. Η χαλάρωση ε, των ε, ε, μέτρων για θεωρήσεις δεν είχε επιπτώσεις πάνω στα αποτελέσματα των εκλογών. Νομίζω ότι αυτά εξαρτήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα ανάμεσα στις 7 και 8 Απριλίου και τις ε, τωρινές εκλογές. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά οι, ε, οι, οι πίκοοι, οι ε, πολίτες συμμετείχαν πολύ περισσότερο στην εκλογική διαδικασία. Για άλλες ερωτήσεις θα ήθελα να πω ότι στα εκλογικά τμήματα είδα άτομα που ερχόντουσαν στα εκλογικά τμήματα και έλεγαν έχετε ένα όνομα στον κατάλογο και αυτό το όνομα δεν διαμένει εκεί ε, που αναγράφεται στον κατάλογο. Δεν ζει ούτε καν στην Μολδόβα και ε, θα ε, ξαναέρθω για να δω αν κάποιος ψήφισε στο όνομα αυτού του ατόμου. Αυτό λοιπόν, αυτή, ε, τα νέα αποτελέσματα οφείλονται σε αυτή τη νέα στάση των πολιτών. Τα εκλογικά τμήματα ήταν καλύτερα οργανωμένα, αλλά υπήρξαν πολλές παρατυπίες, διότι όπως είπα, οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι ακριβής Και υπήρχε ακόμα η δυνατότητα διπλής ε, ψήφου, τριπλής ε, ψήφου ε, λόγω του αριθμού των ταυτοτήτων, των δεχόντουσαν ταυτότητες, διαβατήρια και άλλα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας και κάναμε στην εκθεσή μας μια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε να υπάρξει ε, ηλεκτρονικός εκλογικός κατάλογος, διότι τελειώς δεν θα εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα. Είπαμε επίσης ότι υπήρξαν παρατυπίες, διότι κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας υπήρξαν πολλά προβλήματα, κυρίως ως προς την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση. Όσον αφορά την πολιτική εξέλιξη και την πολιτική κατάσταση αυτή καθεαυτή, υπάρχει μια πλειοψηφία για εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου και αυτό συνέβη. Υπάρχει μια πλειοψηφία για την, ε, για την ε, στο σχηματισμό μια κυβέρνηση, και αυτό θα συμβεί πιθανόν, αλλά η αντιπολίτευση δεν έχει αρκετέ ψήφου για να εκλεγεί ο πρόεδρο τη χώρα. Τι θα συμβεί ε, το ε, ένα, η μία λύση θα ήταν ο Μαριάν Λούπου να εκλεγεί πρόεδρο τη χώρα. αυτό θα ήταν καλό αποτέλεσμα αν μερικοί κομμουνιστέ ψηφίσουν γι' αυτόν. Ή ίσως δεν θα πετύχουν να εκλέξουν πρόεδρο και τότε θα πρέπει να υπάρξουν τρίτες εκλογές το 2010. Θα υπάρξει όμως ένα κοινοβούλιο και μια κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι τις τρίτες αυτές εκλογές. Εγώ προσωπικά ελπίζω, απέφχομαι μια τέτοια κατάσταση αλλά εάν γίνει αυτό νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα κερδίσει το 2010 ακόμα περισσότερες ψήφους από ό,τι τώρα. Ωστόσο, για να αποφύγουμε μια πραγματική πολιτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει σημαντική υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Χαιρετίζω αυτό το πρόγραμμα, το πακέτο των 4 εκατομμυρίων, αλλά η δημοκρατία της Μολδόβας ζει μια βαθιά οικονομική κρίση. Αν δεν τους βοηθήσουμε, κάποιος άλλος θα τους βοηθήσει και τότε θα έχουμε ίσως διαφορετικά εκλογικά αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το ποιο θα τους βοηθήσει, εμείς ή κάποιος άλλος. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινέσκου για την παρέμβασή του αυτή που νομίζω, νομίζω ότι απάντησε διεξοδικά σε όλες τις ε, αντιρρήσεις που προτάχθησαν και ε, αναγνωρίζουμε το ότι υπήρξε μία διεξοδική παρουσίαση. Η παρακάλεσα τον Επίτροπο Όλη Ρεν να καθυστερήσει λίγο, γιατί έφτασε ο Επίτροπος. Α, όχι ακόμα. Μπορούμε λοιπόν να διακόψουμε για πέντε λεπτά. Αλλιώς, ε, α, έρχεται, έρχεται, εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος να διακόψουμε ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή. γιατί καθυστερήσαμε στην ε, αρχή της συνεδρίασης. Ανακτούμε όμως τον ε, χαμένο χρόνο. Eh, Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τη νέα σας ε, ιδιότητα, διότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου ε, έχει αλλάξει η σύνθεση της ομάδας Κατά τους προσεχείς ε, μήνες θα συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να έχετε το χρόνο να εκθέσετε τα ζητήματα που επιθυμείτε. Στις 14 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, θα εγκρίνει το πακέτο της διεύρυνσης. Δηλαδή, θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις στην Κροατία, Μακεδονία, Τουρκία και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Γνωρίζω ότι ο Επίτροπος ε, δέχτηκε να παρουσιάσει αυτό το πακέτο. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων. Στις 15 ε, Ιουλίου η Επιτροπή πρότεινε να μην υπάρχει υποχρέωση ε, θεωρήσεων για τους κατοίκους της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Εμείς ε, ταχθήκαμε υπέρ αυτής της υπόδειξης και χαιρετήσαμε αυτή την παρέμβαση γιατί στο μεταξύ ζητήσαμε την κατάργηση των θεωρήσεων αν και εξαιρέθηκε η Βοσνία Ερσεγοβίνη και η Αλβανία από αυτό το καθεστώς. Ελπίζουμε ότι το στίγμα της Επιτροπής θα οδηγήσει τους Βόσνιους και τους Αλβανούς να προβούν στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αυτές τις εξελίξεις. Ε, αγαπητέ Επίτροπε, θα θέλαμε να μάθουμε εάν προβλέπονται θετικές εξελίξεις με τις δύο αυτές χώρες κατά τη διάρκεια του 2010. Επίσης, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η πρόοδος για την προσχώρηση της ε, Κροατίας και οι προοπτικές κατάληξης αυτών των διαπραγματεύσεων. Επίσης, ως προς τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε σχέση με την κατάσταση της πρώην Ιουκοσλαβίας και την κατάσταση του Κωσυφοπεδίου, όπου δεν προβλέπεται κατάργηση των θεωρήσεων. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, προβεί μία, ε, θα συντάξει μία έκθεση προόδου για να δούμε ποιες, ποιοι είναι οι δεσμοί με αυτή τη χώρα. Θα σταματήσω σε αυτό το σημείο και δίνω το λόγο στον Επίτροπο και θα τον ακούσουμε βεβαίως με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Thank you. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ως Επίτροπος και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να απευθύνω το λόγο στην εκλεκτή επιτροπή σας και πριν υπησέλθω στα θέματα που ε, σκιαγράφησε και ο πρόεδρος προς συζήτηση σήμερα, θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να σας συγχαρώ όλους για την εκλογή ή επανεκλογή σας και επίσης επιθυμώ να συγχαρώ τον αξιότιμο πρόεδρο κύριο Αλμπερτίνη όπως και όλους τους αντιπροέδρους, ε, εισηγητές συντονιστές για την εκλογή σας. Με αυτή την ευκαιρία επιθυμώ επίσης να συγχαρώ τον Πρόεδρο για την ε, ε, ε νίκη την περασμένη Κυριακή στο Σπάδο στο Βέλγιο της Φόρμουλα και βέβαια ο Κίμι Λάκνεν ε, μπορεί, ο συμπατριώτης μου μπορεί επίσης να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Αυτό για μένα κάτι λέει. Ένας πρώην συνάδελφός σας επίσης, ε, ο, συ... ο αντίπαλος του Άρη Βάτανεν, ε, συμμετέσχε στην ομάδα. Ο Ζαντότ, τι έλεγε. Έλεγε, ε, αν θες να κερδίσεις, πάρε Φιλανδό. If you want to win, take a fin. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την νίκη. Αγαπητοί φίλοι, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, γιατί τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι κρίσιμα για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και εσείς θα επομιστείτε σημαντικές ευθύνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε έπαιζε ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής της διεύρυνσης στην Νατιοανατολική Ευρώπη πρόσφατα ε, μέσα από τις εκθέσεις σας, τις συζητήσεις σας ε, τις πολλές ερωτήσεις, επιστολές που απευθύνατε και σε μένα και προς τους συναδέλφους μου. Θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία των προηγουμένων ετών και προσβλέπω στην συνέχιση της στο μέλλον. Ε, θέσατε παράδειγμα δημοκρατικής λογοδοσίας που παραθέτω συχνά στις επαφές που έχω με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ή την Τουρκία δεν θα μπορούσα να ευχηθώ ε, έναν καλύτερο συνεργάτη και εταίρο από αυτή την Επιτροπή. Ας ε, θυμηθούμε λίγο το υπόβαθρο της διεύρυνσης. Ε, πριν από 20 χρόνια, στις 10 Σεπτεμβρίου του 89, η Ουγγαρία πρώτη άνοιξε τα σύνορα με την Αυστρία και επέτρεψε σε χιλιάδες Ανατολικογερμανούς να περάσουν στη Δύση. Αυτές οι εικόνες ε, μας επηρέασαν όλους. Μετά χρειάστηκαν δύο μήνες ακόμη μέχρι να πέσει το τείχος. Το φάρος, ε, η ευτυχία των Ούγγρων ε, βρήκε μιμητές ε, σε άλλες χώρες για να θριαμβεύσει η ελευθερία που οδήγησε στο τέλος του ολοκληρωτισμού. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου, η αρχή ενός δημοκρατικού μετασχηματισμού της Υπήρου μας και αυτό θα πρέπει να μας δώσει τροφή για προβληματισμό και σκέψη. Τώρα, 20 χρόνια αργότερα, είμαστε μια ένωση 27 κρατών μελών που επέλεξαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κήθηκε μια μαγνητική έλξη του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Πρόκειται για μια ένωση που προσφέρει ευημερία, ασφάλεια, αλληλεγγύη ε, και μια σειρά από κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήσαμε την διεύρυνση μέσα από το πρίσμα αυτού ε, του ε, ε, ανοιχτού πνεύματος θέλοντας να θέσουμε ένα τέλος στο, στη διέρεση της Ευρώπης και να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπως ήθελαν οι ιδρυτικοί πατέρες της Ένωσης σήμερα ε, έχουμε τη μεγαλύτερη ε, ε, διεθνή οικονομία, παίζουμε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο αλλά και στην ρύθμιση της πολιτικής διεθνώς. Το η επόμενη πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε τη θέση μας στο μέγιστο βαθμό. Η συνθήκη της Λισαβόνας στην εξωτερική πολιτική σκοπό έχει να ενισχύσει την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε δράση και να ε, είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε να με τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα πιο αποτελεσματικά σε όλο τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι απόλυτα σαφές για μένα ότι η οικονομία και οι θέσεις εργασίας ε, είναι τα πρώτη στα μελήματα ε, των πολιτών μας σήμερα. Είναι πολύ σωστό λοιπόν να βρίσκονται στην, ως πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρώπης και αυτό το ε, είδαμε ε, πρόσφατα και στις εκλογές. Γι' αυτό ε, αρχίσαμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης και γι' αυτό τώρα στο, φροντίζουμε τόσο πολύ την επόμενη Σύνοδο Κορυφής των G20 στο Pittsburgh. Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση όμως δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το σημαντικό έργο της σταθεροποίησης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό να εξαγάγουμε την σταθερότητα στα Βαλκάνια από ότι να εισάγουμε την αστάθεια από εκεί. Σε σύγκριση με πολλές άλλες περιφέρειες στον κόσμο, η Νοτιοανατολική Ευρώπη απολαμβάνει σχετική πολιτική σταθερότητα προς το παρόν ε, μεταξύ άλλων και χάρη στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών εκεί. Αν όμως μας δίδαξε κάτι ο 20ος αιώνας, ε, είναι η ε, ανάγκη να μην είμαστε συγκαταβατικοί προς τα Βαλκάνια. δεν υπάρχει μια αντιστρέψιμη σταθερότητα, ακόμα τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει εφευρεθεί. Υπάρχει και ένας άλλος εξίσου σημαντικός ε, λόγος για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος ε, παίχτης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα που έχουμε να ε, βοηθούμε τις γειτονικέ χώρες. Η ήπια δύναμη της Ευρώπης είναι σημαντικό να ασκηθεί στα Δυτικά Βαλκάνια και από την εργαλειοθήκη της διεύρυνσης και ε, αντλούμε και από την ε, εταιρική σχέση προς τις ε, ανατολικές χώρες. Η ευρωπαϊκή προοπτική για όλες αυτές τις χώρες είναι μια τεράστια υπόσχεση και ένα κίνητρο για τη συνέχιση των δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πιέσαμε πολύ για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, ε, που, ένα θέμα που έθεσε προς συζήτηση σήμερα ο πρόεδρός σας. Γνωρίζομαι πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν θεωρήσεις ε, για τους ε, πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλουμε όλοι να ωφεληθούν από το καθεστώς αυτό, στο βαθμό βέβαια που οι κυβερνήσεις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ε, να εξηγήσω πώς ε, εργαστήκαμε. Κάθε χώρα ε, έλαβε έναν οδικό χάρτη πέρυσι που προδιέγραφε τα προαπαιτούμενα, τα οποία ήταν ασφαλή βιομητρικά διαβατήρια, καλύτερη έλεγχη στα σύνορα, μέχρι ενισχυμένη καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η πρόοδος κάθε χώρας αξιολογείται από τότε ε, ξεχωριστά. Τον Ιούλια προτείναμε να δώσουμε ε, να, στους ε, κατοίκους της Φύρομ, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία ελεύθερη πρόσβαση από τον Ιανουάριο του 2010 να καταργηθούν οι θεωρήσεις δηλαδή από την αρχή του επομένου έτους με την προϋπόθεση ότι το Μαυροβούνιο και η Σερβία ε, θα χρειαστούν κάποια προαπαιτούμενα συγκριτικής αξιολόγησης ακόμη. Ελπίζω ότι η πρότασή μας θα εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως εσείς θα συμμετάσχετε στις διαβουλεύσεις στο θέμα αυτό, υπολογίζοντας την υποστήριξή σας στην πρόταση αυτή. Επίσης, κοινό στόχος είναι η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη να ακολουθήσουν σύντομα τους γείτονές τους. Εάν οι μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν όπως τώρα, ε, τότε η Κομισιόν μπορεί να σκεφτεί ε, να υποβάλει νέα πρόταση στα μέσα του επομένου έτους 2010. Η ταχύτητα της πρόοδου αυτών των χωρών προς ε, την κατάργηση των θεωρήσεων στα ταξίδια είναι στα χέρια των ηθινόντων τους το υπογραμμίζω, η μπάλα είναι στο γήπεδό τους. Όταν ανταποκριθούν στα προαπαιτούμενα θα υποβάλουμε και εμείς νέα πρόταση για τις δύο χώρες. Εν πάση περιπτώσει, όταν τεθεί η πρόταση σε ισχύ, το νέο βιομετρικό διαβατήριο θα είναι αρκετό για να ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σέγγεν και αυτό σημαίνει ότι δεν θα ε, συνοστίζονται στις πρεσβείες, δεν θα πληρώνουν για τις θεωρήσεις, δεν θα πρέπει να ε, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά και οι πολίτες των χωρών αυτών θα μπορούν να επισκέπτονται οικογένειες και φίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειάζονται να μπαίνουν σε αυτές τις επίπονες ε, διαδικασίες διέλευσης και θα είναι δυνατόν οι νέοι να σπουδάζουν στις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της Ένωσης. Ε, με δύο λόγια αυτό σημαίνει μια ε, ένα περαιτέρω εξευρωπαϊσμό της κοινωνίας των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό δείχνει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι μόνο ένα θέμα ολοκλήρωσης ε, εθνών, αλλά και λαών και πολιτών. Αυτό είναι ο αρχικός και θεμελιώδης στόχος μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πριν ε, τελειώσω θα ήθελα να σας παρουσιάσω την παρούσα κατάσταση με τις χώρες της διεύρυνσης. Για την Κροατία. Αν η Κροατία ε, πληρεί ε, πληρώσει έγκαιρα τα benchmarks, τα πρωτοπετούμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την δικαστική εξουσία και τη συνεργασία και αν ε, λυθεί το θέμα των συνόρων με τη Σλοβενία θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις προσχώρησης κατά το πρώτο εξάμεινο του επομένου έτους. Εγώ ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο και σημειώνω ότι υπάρχει ε, σημαντική βελτίωση στην πολιτική ατμόσφαιρα, στο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών και των ηγετών τους τώρα και αυτό νομίζω ότι δικαιολογεί κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία εις ό,τι αφορά την διευθέτηση του συνοριακού προβλήματος Κροατίας-Σλοβενίας σύντομα. Επίσης ελπίζω να ξαναρχίσουν στην Τουρκία βασικές μεταρρυθμίσεις ε, την επόμενη περίοδο, επειδή η πρόοδο τη διαπραγματεύσεις προσχώρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που θα γίνει στις νομοθετικέ μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, ε, ε, θρησκευτικέ ελευθερίε, ελευθερίες, ελευθερία έκφρασης, δικαιώματα μειονοτήτων, συνδικάτων κλπ. Χαιρετίζουμε επίσης τις πρόσφατες διαβουλεύσεις ε, σε ό,τι αφορά μια κουρδική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία για το κουρδικό, που ελπίζομαι ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις για να ε, βελτιωθούν τα ε, γλωσσικά και θρησκευτικά δικαιώματα όλων των Τούρκων ε, αλλά και μια ανάπτυξη στη νοτιοανατολική Τουρκία και ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα παίξει επικοδομητικό ρόλο στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού και τη βελτίωση του πολιτικού κλίματος αν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πληρώσει τα benchmarks που απαιτούνται, η Κομισιόν θα μπορέσει να προτείνει φέτος να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις προσχώρησης επίσης. Το όνομα δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά είναι σαφές ότι μία λύση του προβλήματος αυτού θα δημιουργούσε πολύ θετικότερο κλίμα και περιβάλλον για την συνέχιση της διαδικασίας προσχώρησης. Το Μαυροβούνιο συνεχίζει να δίνει καλά, καλές ειδήσει. Ε, βλέπουμε πάνω εκεί τι μπορεί να επιτευχθεί αν υπάρχει εθνική συνένεση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αν τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό πρόγραμμα. Ε, τώρα ε, σε λίγου μήνε θα προετοιμαστεί η γνωμοδότηση τη Επιτροπής ε, για τη χώρα αυτή. Οι πρόσφατε εκλογές στην Αλβανία ε, έλαβαν χώρα με καλύτερες προϋποθέσεις ε, από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αν και υπάρχουν ακόμα δυναμίες. θέλουμε να το, και ο ΑΣΕ να αποφανθεί οριστικά μετά πάνω στη διεξαγωγή των εκλογών. Η Κομισιόν θα ετοιμάσει τη γνωμοδότηση για την Αλβανία όταν το ζητήσει το Συμβούλιο. Μετά, η Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Ε, είπα πολλές φορές στους ηγέτες ε, της χώρας ε, ότι το 2009 θα μπορούσε να αποβεί κρίσιμο έτος για τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Ακόμα πληρούν, μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τις την απαλλαγή από τις θεωρήσεις το 2010. Επίσης πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετάβαση προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δηλαδή το γραφείο του ΙΠΑ του εκπροσώπου να κλείσει και να μπορεί ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία εκεί. Αυτό θα ανοίξει την πόρτα για ε, υποψηφιότητα για ένταξη και θα αποτελέσει μια μεγάλη, μια τεράστια ευκαιρία για αυτή τη χώρα. Όμως, δυστυχώς, προς το παρόν δεν βλέπω η ηγεσία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να δίνει δείγματα γραφής που θα μας οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν η Βοσνία Ερζεγοβίνη θα χρειαστεί πολύ προσοχή ε, και στρατηγικό σχεδιασμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, από την πλευρά τη δική σας, από την πλευρά του Συμβουλίου ε, και από τους διεθνείς εταίρους μας. Στη Σερβία η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για τις μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα ε, ε, εφαρμόζουν την προσωρινή συμφωνία σε μονομερή βάση παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας και έτσι επιδεικνύουν, αν θέλετε, την ισχυρή ευρωπαϊκή βούλησή τους. Επίσης, ε, πραγματοποιείται το πρόγραμμα ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης αποτελεσματικά. Ε, ασχολούνται με σοβαρότητα με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τον οδικό χάρτη για τις θεωρήσεις και έχουν έχουν ε, πρόσφατα επιτύχει ε, μεγάλες βελτιώσεις. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει την πρόοδο της Σερβίας ε, και να ξεμπλοκάρει η προσωρινή συμφωνία. Το κοσυφοπέδιο είναι σταθερό αλλά εύθραυστο. Το νομικό πλαίσιο εξελίσσεται, η εφαρμογή του λιγότερο καλά. Ε, υπάρχει θέμα κράτους δικαίου ε, δικαστικής εξουσίας. Τον Οκτώβριο, στα πλαίσια του πακέτου διεύρυνσης, στα μέσα Οκτωβρίου, θα αξιολογήσουμε το τι πρέπει να κάνει το κοσυφοπαίδιο για να ανταποκριθεί στην ευρωπαϊκή του προοπτική. Κρίσιμα θέματα της μελέτης είναι οι επαφές ε, μεταξύ των κοινοτήτων, των ανθρώπων, κινητικότητα, εμπόριο, περιφερειακή συνεργασία. Για την Κύπρο. Οι συνομιλίες ε, Χριστόφια Ταλάτ μπαίνουν σε αποφασιστική φάση. Ε, γίνονται διαπραγματεύσεις με πολύ δούνε και λαβίν. Πρέπει να ε, αρχίσουν πάλι αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω ότι φέτος και του χρόνου θα δούμε να λύνεται το πρόβλημα, να ενοποιείται η Κύπρος και ο κύριος Μπαρόζο θα συμβάλλει και εκείνος κατά το δυνατόν ε, στην επίσπευση της επίλυσης. Ε, για την Ισλανδία τέλος, η Ισλανδία είναι ευρωπαϊκή χώρα με μακρές και βαθιές ευρωπαϊκές ρίζες, δημοκρατικές ρίζες και ήδη μέσα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ε, και τη συμμετοχή στο χώρο του Σέγγεν ε, συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ήδη κατά δύο τρίτα εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο. Όμως δεν υπάρχει ταχεία διαδικασία για την Ισλανδία, δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να ε, περικοπεί η διαδρομή μέχρι την ε, ένταξη. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί η χώρα αυτή είναι παρόμοια με όλες τις υποψήφιες χώρες ε, και θα κρυθούν και θα κρυθεί και αυτή η χώρα χωριστά. Θα πρέπει η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει για τη γνωμοδότησή της την ίδια μεθοδολογία όπως και για τις άλλες υποψήφιες χώρες. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, για να ε, ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να αναφερθώ στις κοινοβουλευτικές ακροάσεις ε, πριν από πέντε χρόνια, σχεδόν ε, ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, ε, όταν ε, κατά στην ακρόαση ε, ερωτήθην για το πρόγραμμα της διεύρυνσης στην επόμενη πενταετία. Είπα ότι εγώ ήθελα να κάνω τη δική μου τη δουλειά σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πάνω σε έξι στόχους που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι το 2009, το τέλος του 2009. Πρώτον, το 2009 θα έπρεπε να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών. Δεύτερον, η διαδικασία ε, ένταξης της Κροατίας θα έπρεπε να φτάσει στο, στην κατάληξή της. Ε, τρίτον, οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα έπρεπε να ε, έχουν πια σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό μέσα από συμφωνίες σύνδεσης. Τέταρτον, η Τουρκία θα έπρεπε να είναι σταθερά σε μια ευρωπαϊκή τροχιά. Πέμπτον, το καθεστώς του κοσυφοπεδίου θα έπρεπε να έχει διευθετηθεί και έκτον θα έπρεπε να ενοποιηθεί ε, η Κύπρος. Ε, πέντε από τους έξι στόχους ε, έχουν πληρωθεί, όχι τέλεια, όχι 100% αλλά έχουμε φτάσει εκεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα παραμένουν σοβαρές προκλήσεις και διμερεί θέματα που έχουν τώρα καταστεί ευρωπαϊκά προβλήματα. Αγαπητοί φίλοι, ε, σήμερα ε, η Ευρώπη έχει ενοποιηθεί πάλι, είναι ελεύθερη. Ας παραμείνει έτσι. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη το έργο μας, όπως και στη Βόρειο Ευρώπη. Είναι δύσκολη αποστολή, αλλά πολύ σημαντική. Εσείς θα παίξετε ρόλο κέριο για να γίνουν όλα αυτά, για να έχουμε επιτυχία και εύχομαι στις εργασίες σας και στην αποστολή σας κάθε επιτυχία. Ε, εύχομαι καλή συνεργασία μεταξύ ημών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τη σαφή του εισήγηση. Τώρα μπαίνουμε στη συζήτηση. Έχω 27 συναδέλφους που ζητούν το λόγο, άρα δεν μπορώ να δεχτώ άλλες παρεμβάσεις εκτός από αυτές που έχουν καταγραφεί. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές όχι περισσότερο από 1,5 λεπτό όπως ίσχυσε και σήμερα το πρωί. Ζήτω συγγνώμη εκ των προτέρων για αυτό το περιορισμό, αλλά είναι αναγκαίος για οργανωτικούς λόγους. Ο κύριος Σαλαφράνκα για 1,5 λεπτό. επειδή λίγη η θητεία της Επιτροπής θα πρέπει να φτάσουμε σε έναν απολογισμό δραστηριοτήτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όλι Ρεν για την εργασία του, το έργο του γενικότερα. Επίσης θα ήθελα να του διατυπώσω ορισμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ως προς την Ισλανδία. Υπάρχει ένα fast track όπως ξέρετε υπάρχει, ε, είχαμε ε, μία πολύ ε, σχετική πλειοψηφία και σε σχέση με τις διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας και Αρμηνίας. Πώς προβλέπεται η κατάσταση την επόμενη εβδομάδα. Επίσης έγινε λόγος για την λήξη των διαπραγματεύσεων με την Κροατία σε έξι μήνες. πιστεύετε ότι σε αυτή την προθεσμία θα έχει ε, επιληθεί η διαφωνία που υπάρχει μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και το καθεστώς των θεωρήσεων. τον Ιούλιο η Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτική βοήθεια για την Σερβία, Τουρκία και άλλες χώρες των Δυτικών, Αλφα, ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Σαλαφράνκα. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Βίγκενιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Δεν θα ήμουν ε, μέλος ε, αυτού του κοινοβουλίου αν δεν είχατε επιτύχει με τη διεύρυνση με τη χώρα μου. Θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθεροποίηση του καθεστώτος των θεωρήσεων αυτή την απόφαση για να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα οι κάτοικοι της Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία διότι είναι ένα βήμα για την προσχώρηση των χωρών αυτών. Υπάρχει όμως ένταση διότι η Αλβανία και η Βοσνία Αρζεγοβίνη δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο. Νομίζουμε ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ποια είναι τα προβλήματα της Αλβανίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης τα οποία παρεμποδίζουν ε, την, ε, την συμπερίληψή τους ε, στο πακέτο αυτό. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για την κατάσταση με την Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου υπάρχουν πάρα πολλοί υπήκοοι της Σερβίας που έχουν διπλή ηθαγένεια και που θέλουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόσφατα, ο, στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργό Ερντογάν στην επίσκεψή του εδώ μίλησε για την Τουρκία, για τις ελπίδες της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσανατολισμό. Είναι μήπως ε, η Τουρκία ε, πλησιάζει την Ευρώπη. Η κυρία Νέιτς έχει τον λόγο. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε στο χρόνο που έχετε. Ε, θα ευχαριστώ ε, τον Πρόεδρο και τον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάντοτε όταν βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή μας και εξ ονόματος της ομάδος μου θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλη την καλή δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα και που θα συνεχίσετε να κάνετε. Στις ερωτήσεις μου θα ήθελα να εστιαστώ στην εξαίρεση για τις θεωρήσεις, την παρέκκληση. Χαίρομαι που οι κάτοικοι του Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας από την 1η Ιανουαρίου δεν θα χρειάζονται θεωρήσεις για να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αλλά όπως και οι προλαλήσοντες λυπούμε ότι αυτό δεν θα καταστεί δυνατόν για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Δεν θα μπορούσαμε, κύριε Επίτροπε, να πούμε ότι αν οι χώρες αυτές υιοθετούσαν το ένα ή το άλλο μέτρο, τότε ε, οι υπήκοοι τους θα μπορούσαν να επιτύχουν αυτήν την εξαίρεση από θεωρήσεις. Νομίζω ότι όσον αφορά στην ποσνια Ριζεγοβίνη, αν η κατάσταση διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, τότε οι ε, Σέρβοι της Βοσνίας και οι Σέρβοι της Κροατίας θα προσπαθήσουν να επιτύχουν διαβατήρια στις χώρες αυτές και η τάση αυτή θα βαίνει αυξανόμενη. Δεν μας είπατε τίποτα για τις παρεκκλήσεις, αποθεωρήσεις για το κοσυφοπέδιο. Ξέρω ότι το θέμα είναι πολύ λεπτό, αλλά θα ήθελα να έχω την δική σας άποψη ως προς το θέμα αυτό. Τώρα δίνω τον λόγο ε, στον κύριο Λούνατσεκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτρο Περέν, ευχαριστώ για την πολλή δουλειά που κάνει η Κομισιόν για τη διεύρυνση. Και εγώ θέλω να μιλήσω για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και να κάνω και μια άλλη ερώτηση για το Κωσίφο πέδιο και μετά για την Τουρκία. Καταρχήν, απελευθέρωσαν θεωρήσεων. Συμφωνώ με αυτό που είπε πριν από λίγο η συνάδελφο Νίτσε και για μας και για την ομάδα των Πρασίνων. Ε, είναι σημαντική η μεγαλύτερη ελευθερία στις ε, θεωρήσεις και στο ε, Μαυροβούνιο κλπ. Αλλά στη Βοσνία μπαίνει το θέμα και για την Αλβανία υπάρχει ζήτημα. Και τίθεται το ερώτημα και με τη Σερβία, το είπατε και εσεί. η Σερβία πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Και αυτό που κατάλαβα και από τι συνομιλίε και από τον τύπο, τα μέσα ενημέρωση είναι ότι ήταν πολιτική απόφαση αυτό ε, από την πλευρά της Σερβίας. Ε, γιατί δεν, χρειάζεται, δεν μπορούμε και για τη Βοσνία να το πούμε αυτό ε, με τη για ότι νιώθουν οι μουσουλμάνοι Βόσνοι αποκλεισμένοι. Γιατί δεν είναι δυνατόν και για τη Βοσνία να μιλήσουμε για πολιτική απόφαση και ότι θα υπάρξει αυτή η απελευθέρωση. Είπατε επίσης ότι η Κομισιόν στα μέσα του 2010 θα υποβάλει νέα πρόταση. Είχα ε, θεωρήσει ότι αυτή η απόφαση θα λαμβάνεται ήδη τον Νοέμβριο, νωρίτερα δηλαδή θα, κάναμε, ε, θα δίναμε μια όθηση. Επίσης, ε, ήρθε χθε ο Πίτερ Φέιθ να μας μιλήσει για το κοσυφοπαίδιο, ε, για τις ε, ε, δημοτικές εκλογές. Υπάρχει μια υποστήριξη από την πλευρά της Κομισιόν των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Σερβία που για τους Σέρβους, που θέλουν να προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν τους Σέρβους, Κωσοβάρους για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Ο κύριος Τάνοκ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρεν. Καλώς ήρθατε ε, στην ε, Επιτροπή μας. Ε, είμαστε υπέρ της διεύρυνσης, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης θα πρέπει να πληρούνται 100% πριν προσχωρήσουν νέες χώρες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης το γεγονός ότι η κόποση της διεύρυνσης από την κοινή γνώμη είναι έντονη και θα πρέπει να τους πείσουμε για τις αρετές της διεύρυνσης, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την Ισλανδία είναι ιδιαίτερη περίπτωση περίπτωση ε, λόγω του καθεστώτος του, της χώρας και της μικρής οικονομίας. Έτσι λοιπόν καλό θα ήταν να υπάρχει ένα fast tracking, μια συνοπτική διαδικασία για τα Δυτικά Βαλκάνια, μεγαλύτερη διπλωματική πρόκληση. Χαιρετίζουμε το έργο σας. Μας ενδιαφέρει βέβαια η σταθερότητα πολιτική στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, προβλήματα διαφορά οργανωμένου εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαι ιδιαίτερο φίλος της Μακεδονίας, ελπίζω ότι θα αρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Τέλος χαιρετίζω αυτό που είπατε για την Κύπρο, μια χώρα ιδιαίτερα αγαπητή. Για μένα ε, πάντοτε ε, είμαστε υπέρ της αξιοποίησης κάθε δυνατότητας υπό την αιγίδα και των Ηνωμένων Εθνών, αλλά υπάρχει και η Τουρκία ως τρίτος, ε, τρίτο μέλος. Και ελπίζω να ασκήσετε την επιρροή σας στην Τουρκία, ούτως ώστε να ε, φροντίσετε για επιτυχία έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο. Ο, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Όλη Ρεν για τη δουλειά που κάνει μέχρι στιγμής. Εμείς σαν εκπρόσωποι εδώ και της Κύπρου θέλω να διαβεβαιώσω ότι είμαστε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα των 100 εκατομμυρίων. Είμαστε υπέρ της ένταξής της, θα τολμούσα να πω ότι θέλουμε να γίνουμε και το όχημα για να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον βέβαια υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον πράγματι δουλέψει επικοδομητικά για τη λύση του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρότυπο κάθε προηγούμενης ενταξιακής διαδικασίας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων από μέρους της Τουρκίας η οποία δυστυχώς συνεχίζει να μην εφαρμόζει το πρωτόκολλο της Άγκυρας που υπέγραψε και κρατά κλειστά λιμάνια και αεροδρόμια σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα. Εμείς κύριε Όλη Ρεν δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε ένα πρόβλημα. Εμείς θέλουμε και προσπαθούμε να λύσουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι χωρίς λύση στο Κυπριακό, με απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, με αναχέτηση της θέλησης της Τουρκίας να αποτελεί και μετά την λύση εγκύτρια δύναμη της δημοκρατίας της Κύπρου ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μη λύσης τότε η Κύπρος και δεν το λέω αυτό καθόλου για εκβιασμό τότε η Κύπρος θα είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί στη λύση του Κυπριακού. Θέλουμε να ακούσουμε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, τι είναι αυτό που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. La parola all'onorevole Belder. Raccomando... Belder, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο του 1,5 λεπτού. Dank u Κύριε Επίτροπε, eh, eh, eh, σας ευχαριστώ ε, και θα ήθελα να δούμε το σοβαρό θέμα στην Τουρκία. Σήμερα χριστιανοί εθελοντές βρίσκουν τις πόρτες κλειστές ε, στα ε, γυροκομεία για τους γέρους. Μετά από χρόνια σχέσεων χωρίς προβλήματα υπάρχει τώρα μια άρνηση ε, για τους, αυτούς τους χριστιανούς και φοβούνται οι χριστιανοί ότι επειδή είναι χριστιανοί δεν θα μπορούν πια να επιτύχουν τη βοήθεια από τα ιδρύματα αυτά στην Τουρκία. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να ζητήσετε διευκρινήσεις από τις τουρκικές αρχές, ούτως ώστε η κατάσταση αυτή να μην υπάρχει πια, να τεθεί τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Θα θέλαμε μια απάντηση για το θέμα αυτό. Σας εύχομαι καλή τύχη στη δουλειά σας. Ο κύριος Μπάρτλενερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάνατε καταστροφική δουλειά αυτήν ε, τα τελευταία χρόνια ε, για τους πολίτες ε, του Ολλανδούς ήταν κακά τα πράγματα για, με τη Ρουμανία και την Βουλγαρία διότι στην Ολλανδία υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση λόγω των εγκληματιών που έρχονται από τις χώρες αυτές και εσείς ο ίδιος ομολογήσατε την αποτυχία σας αλλά συνεχίζετε αυτή την κακή δουλειά πρέπει να σταματήσετε την αυτήν ε, την δουλειά της διεύρυνση. Δεν χρειαζόμαστε την Τουρκία, την Αλβανία, την Βοσνία. Ο εξισλαμισμός της Ευρώπης είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Μπορεί οι χώρες αυτές να είναι καλοί γείτονε, αλλά δεν πρέπει να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και αν ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις θα έχουμε περισσότερους εγκληματίες και τρομοκράτες στη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι για τη Βοσνία δεν θα υπάρχουν θεωρήσεις θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους Ολλανδούς ε, πολίτες είσαστε μεγαλομανείς. Σταματήστε τον εξισλαμισμό της Ευρώπης και να γυρίστε στη χώρα σας και να μην ξανάρθετε ποτέ εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Αλλά παρόλα, la collega Omen Reuten. Omen Reuten. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά για μένα μετά τον αγαπητό συνάδελφο Μάντλενερ που μόλις εξελέγει που μπορώ να λάβω τον λόγο σε αυτό το κοινοβούλιο και να μιλήσω ε, για τη διεύρυνση με τρόπο τελείως αντίθετο με τα όσα λέχθηκαν. Έχω μεγάλο σεβασμό ε, για τη δουλειά ε, του Επιτρόπου για το πώς αντιμετώπισε το φάκελο της διεύρυνσης. Ξέρουμε όλοι, όλοι πολύ καλά ότι επειδή είμαστε δημοκράτες ότι έγιναν διάφορα σφάλματα αλλά όταν έχουν γίνει σφάλματα όλοι μαζί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διορθώσουμε τα πράγματα. Υποστηρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, και με ε, συγχωρώ που με συγχωρείτε ε, που ξεπερνώ το χρόνο μου, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ειρήνη και ε, την σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως όλοι μαζί. Θέλω να το πω στον κύριο Μάντλενερ ότι παρότι από το 1991. Δεν έχουμε πια το σύμφωνο της Βαρσοβίας χάρη σε αυτή τη διεύρυνση. Εμείς στις κατοχώρες είμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε όλοι σε καλύτερη κατάσταση. Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Και τώρα όσον αφορά στην Τουρκία και την Αρμενία, αυτή η προσέγγιση είναι θετική είναι επίσης θετική για την εξέλιξη στο Νότιο Κάφκασο. Είναι επίσης καλή, καλή για τους Κούρδους. Θετική η κατάσταση αυτή, ε, διότι η νομοθεσία έχει βελτιωθεί και θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτω ώστε να μεριμνήσουμε να συνεχιστεί αυτή η καλή εξέλιξη. Μπορούν να γίνουν πολλά καλά πράγματα υπάρχουν ε, οι αποφάσεις του ποινικού δικαστηρίου κλπ. κλπ. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να έχουμε μια καλύτερη συνεννόηση με την Τουρκία για αυτά τα θέματα. Τελευταία παρέμβαση, ε, κυρία Κοπά. Τελευταία χρόνια όλες οι εκθέσεις προόδου για την Τουρκία παρουσιάζουν ένα γενικά θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Σήμερα δυστυχώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Χθε μόλι τουρκικό μαχητικό F-16 παρενόχλησε πολιτική πτήση τη Ολυμπιακή Αεροπορία ενώ προχθές έλαβε χώρα εικονικός βομβαρδισμός πάνω από το ελληνικό νησί Φούρνη. Από την αρχή του 2009 παρακολουθούμε συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι τουρκικά μαχητικά εκτελούσαν χαμηλές υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παραβιάζοντας και το μορατόριο για ε, πάυση στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Τουρκία παράλληλα αρνείται να εφαρμόσει τις συμφωνίες που υπέγραψε με την Ελλάδα το 2002 για υπανεσδοχή παράνομων μεταναστών, αρνούμενη επίσης να υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που έχουμε θετικές εξελίξεις, όπως το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας, την ώρα που ο Πρωθυπουργό Ερντογάν δηλώνει ότι επιθυμεί και το πιστεύουμε ότι εννοεί ειλικρινά να επιλύσει το κουρδικό πρόβλημα, η χώρα αυτή διατηρεί το κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας. Κύριε Επίτροπε, θέλω να τονίσω ότι στην περσινή έκθεση δεν υπήρχε δυστυχώ καμιά αναφορά για το πρωτόκολλο επανεισδοχή. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει πρόθεση να συμπεριληφθεί. Σκοπεύει η Επιτροπή να στυλιτεύσει την επιθετική στάση υποψήφια χώρα προ κράτο μέλο. Θα το συζητήσετε με τι τουρκικέ αρχέ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνοψίσετε, διότι υποβλήθηκε ε, σωρία ερωτήσεων. Θα ήθελα όμως να είσαστε όσο δυνατόν πιο συνοπτικό. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής για τις ε, πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται πιο συνεκτικά για να έχω την ευκαιρία να ακούσω περισσότερα από εσάς. Εκτιμώ πολύ αυτό το διάλογο και αυτή τη συζήτηση μεταξύ μας. Τώρα, σχετικά με το γενικότερο ύφος των ερωτήσεων, μια παρατήρηση, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ε, αφενός έχουμε το θέμα των μουσουλμάνων σε σχέση με την απελευθέρωση των θεωρήσεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και παράλληλα ε, ε, δουλεύομαι υπέρ της ε, βελτίωσης της διακίνησης των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Προσπαθώ να δω κάθε χώρα και το, τα δεδομένα που υπάρχουν, να τα εκτιμήσω χωριστά και αυτό είναι μια πολιτική που είχε βρει σύμφωνο και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ε, για την αξιολόγηση κάθε χώρας, ούτως ώστε να σημειωθεί η πρόοδος αμέσως μόλις ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέσαμε. Ε, δεν ε, έχω πρόβλημα να ξαναγυρίσω στη Φιλανδία. Ήταν εξαιρετική, εξαιρετικό το καλοκαίρι και λόγω της αλλαγής του κλίματος. Αλλά ε, ναι, ευχαρίστω να ξαναγύρισα εκεί. Αλλά δεν έχω αναλάβει ορισμένε υποχρεώσει στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεν θέλω να πάρω ένα εισιτήριο χωρί επιστροφή προ την ε, Φιλανδία πάλι. Τώρα, ε, για τι ερωτήσει των ε, αρκετών βουλευτών και την κυρία, της κυρία και την κυρία Νάιτ και άλλων, θα ήθελα να σας πω τους λόγους για τους οποίους η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν συμπεριελήφθησαν στην τωρινή πρόταση που υποβάλαμε τον Ιούλιο για ε, απαλλαγή από τις θεωρήσεις ε, στα ταξίδια ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο λόγος είναι απλός. Η χορήγηση απαλλαγής θεώρησης για πολίτες ιασδήποτε χώρας δεν είναι θέμα μιας και μόνο πολιτικής απόφασης. Έχει σχέση με τις προϋποθέσεις, τους όρους που πολλές φορές είναι τεχνικής φύσεως, αλλά παρόλα αυτά είναι ουσιώδης και πρέπει να πληρούνται. Είναι αναγκαίο αυτό. Ο χώρος του Σένιν είναι κοινό χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας διακίνησης ανθρώπων 28 κρατών προς το παρόν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών που διαβιούν σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας βέβαια. Ε, υπάρχουν υψίστα ε, κριτήρια ασφαλείας που πρέπει να ισχύουν στα εξωτερικά σύνορα του χώρου του Σένιεν. Γι' αυτό και μόνο η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, τον Ιούλιο δεν, ήταν, δεν θεωρήθηκαν ακόμη όριμες για να συμπεριληφθούν στην πρότασή μας. Και μάλιστα εφαρμόζομαι την λογική που εξέφρασε η κυρία Νάιτς, γιατί είπατε γιατί δεν φροντίζεται ώστε αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι χώρες να αποτελέσουν ε, μέρος των προτάσεων. Με αυτό κάναμε. Με άλλα λόγια, όταν ε, μπορέσουν να μας πείσουν ότι βραχυπρόθεσμα θα είναι σε θέση να πληρούν τις προϋποθέσεις. Μόλις αυτό γίνει, μόλις πληρούν τις προϋποθέσεις, θα κάνουμε και την πρόταση. Ο χρονικός ορίζον ε, θα είναι τέτοιος ώστε οι χώρες αυτές να επιτύχουν το στόχο τους ε, από τα μέσα του επομένου έτους του 2010 υπό την προϋπόθεση, υπό τον όρο ότι θα πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα. Ποια είναι τα εκκρεμή θέματα για την Αλβανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι η ευρεία εισαγωγή βιομετρικών διαβατηρίων, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και εφαρμογή των πολιτικών αυτών στην πράξη, επίσης ενίσχυση συνοριακών ελέγχων και διαχείρισης ε, της μετανάστευσης. Είναι καθήκον μου, καθήκον μας και το καθήκον του Αντιπροέδρου του Ζακ Μπαρό και όλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πείσουμε όλους τους ε, υπουργούς εσωτερικών των κρατών μελών μας ότι οι χώρες για τις οποίες συζητούμε έκαναν αυτό που έπρεπε σε αυτό το τομέα. Πρέπει να επαγρυπνούμε και πρέπει να είμαστε και αυστηροί στις αναλύσεις και εκτιμήσεις μας. Υπάρχει επιστολή που αναφέρει τους συγκεκριμένους τομείς για τους οποίους, στους οποίους, για παράδειγμα, η Βοσνία Ζεγοβίνη καλείται να επιτύχει μεγαλύτερη πρόοδο ε, στην επιστολή στους υπουργού υπεύθυνου για θέματα ασφάλειας. Και υπάρχουν κάποια σημαντικά παραδείγματα εδώ. Το πρώτο ζήτημα είναι η έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων σε ευρεία κλίμακα. Ε, ένα νέο κεντρικό σύστημα εφαρμόστηκε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη τώρα μόλις, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, δηλαδή μετά την υποβολή της πρότασής μας. Η έκδοση διαβατηρίων βιομετρικών υποτίθεται ότι θα αρχίσει τον Οκτώβριο. Από την άλλη πλευρά, η Φύρομ, Σέρβια και Μαυροβούνιο βρίσκονται ε, σε αυτή την κατάσταση. Πάνω από 420.000 βιομετρικά, διαβατήρια έχουν εκδοθεί στην Φιρόμ. Στη Σερβία πάνω από 700.000 βιομετρικά διαβατήρια. Στο Μαυροβούνιο πάνω από 100.000. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, είναι σημαντικό να πληρούνται κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις τεχνικής φύσεως και όταν αυτό συμβεί εμείς θα προχωρήσουμε και θα υποβάλλουμε την σύσταση που άλλωστε ε, έχουμε ε, υποβάλει για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Για τα άλλα θέματα, σύντομα, για να ε, μας μείνει χρόνος για να συνεχίσουμε τον διάλογο. Για την Ισλανδία, θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος να περιγραφεί η κατάσταση στην Ισλανδία σήμερα σε σύγκριση με άλλες υποψήφιες και πιθανώς υποψήφιες χώρες είναι ότι χάρη στις ε, μακρές βαθιές δημοκρατικές ρίζες της και τη συμμετοχή στον οικονομικό χώρο και τον χώρο του Σέγγεν, ενώ μία άλλη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων είναι στα μισά του δρόμου περίπου, σε αυτό το μαραθώνιο μέχρι την ένταξη, η Κροατία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, αλλά μια ε, χαρακτηριστική χώρα, ο μέσος όρος, είναι στο μέσον του δρόμου. Η, η Ισλανδία είναι ε, στα τελευταία 35 με 40 χιλιόμετρα γιατί, του μαραθωνίου γιατί ήδη έχει, ε, εφαρμόζει τα δύο τρίτα του κοινοτικού κεκτημένου. Βέβαια, οι μαραθωνοδρόμοι λένε ότι μετά το 35ο χιλιόμετρο δυσκολεύουν πολύ περισσότερο τα πράγματα μέχρι τον τερματισμό. Δεν σημαίνει λοιπόν, δηλαδή ότι οι προκλήσεις της Ισλανδίας ε, είναι λίγες, έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει η Ισλανδία. Και τώρα στο τέλος πολύ περισσότεροι από άλλοι. Για ε, τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας, ένα θέμα που... Ε, ανάφεραν η ε, κυρία Κοπά, η κυρία Όμεν μεταξύ άλλων. Ε, υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις και τους τελευταίους μήνες ενθαρρύναμε και την Τουρκία και την Αρμενία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, να αρχίσουν διπλωματικές σχέσεις, γιατί αυτό έχει μεγάλη και θετική επίπτωση στη σταθερότητα της περιοχής του, του Καυκάσου. Τώρα, θέματα που αφορούν την Τουρκία, που ετέθησαν από πολλούς ε, προβουλευτές, τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον κύριο Τάνοκ, τον κύριο Μπέλντερ, την κυρία Ομενρόιτεν, την κυρία Κοπά. Θα ήθελα να αναφέρω αυτό που είπε η κυρία Όμεν για τη σημασία της διεύρυνσης γενικότερα και την διαδικασία προσχώρησης ε, της Τουρκίας ειδικότερα. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι αλλά και σταθεροί με την Τουρκία. Δίκαιοι ε, δηλαδή τηρώντα τι υποσχέσεις μας, τις δεσμεύσεις μας, ούτω ώστε να έχουμε την απαραίτητη βάση για να ζητούμε από την Τουρκία να επιτελέσει πρόοδο πληρώντας τι προϋποθέσεις για την ένταξη. Αυτό είναι ένα ταξίδι, ε, όπου το, το ταξίδι είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με τον προορισμό δηλαδή ε, μεταρρυθμίσεις που ε, είναι, ενισχύουν θρησκευτικές ελευθερίες, άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως είπε ο κ. Μπέλντερ, ελευθερία της έκφρασης, που θα βοηθήσει πολύ στις διαβουλεύσεις και σε όλη τη συζήτηση για την πρωτοβουλία για το κουρδικό, ώστε η Τουρκία να γίνει καλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια των διμερών μας σχέσεων και σε ό,τι αφορά ε, το χειρισμό τεράστιων ε, προκλήσεων όπως η βελτίωση της σταθερότητας ε, στην περιοχή του Καυκάσου ή την διαδικασία την ειρηνευτική στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί διευρύνατε το θέμα. Ο δεύτερος γύρος θα αφορά παρεμβάσεις ενός λεπτού. Γι' αυτό θα ήθελα να διατυπώσετε άμεσα την ερώτησή σας και να είναι μόνο μία. Η κυρία Πακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα. Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, δεν μπορείτε να τα πείτε και όλα και σε ορισμένα ζητήματα δεν μπήκατε στο απαραίτητο βάθος. Είναι σημαντικό για μένα να ξέρω τι σημαίνει όταν λέτε ότι η Κροατία ε, στα μέσα του επόμενου έτους θα περάσουν στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Πότε θα ανοίξουν τα ε, υπόλοιπα κεφάλαια. Είναι δυνατόν αυτό τώρα. Τι θα γίνει με τη Μακεδονία. Λέτε του χρόνου μπορεί. Η Ελλάδα θα συνενέσει αφού δεν θα έχει επιληθεί ενδεχομένως το ζήτημα του ονόματος να προχωρήσουν όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι. Επίσης με τη Σερβία σε ποιο βαθμό ε, έχει ευοδοθεί συνεργασία με το δικαστήριο στη Χάγη. Τέταρτον, κοσυφοπέδιο. Τι γίνεται εκεί. Μεγάλες εντάσεις. Μιλήσαμε τον κύριο Φάιτ χθε και δεν μας είπε τίποτε. Γιατί πρόκειται για το θέμα της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και EULEX. Εκεί η EULEX δεν κάνει υπέρβαση, αν θέλετε, καθηκόντων και ενδεχομένως δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια στο κοσυφοπέδιο που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε ταραχές στο δρόμο. Ε, τι λέτε πάνω σε όλα αυτά. Ο κύριος Βόμποτα έχει το λόγο. Καμία εισαγωγή σας παρακαλώ να υποβάλλετε μία ερώτηση και μόνο. Thank uh, Ευχαριστώ. Στο θέμα των θεωρήσεων ε, λυπούμε για την κατάσταση, αλλά κατανοώ τα επιχειρήματά σας, τα οποία και υποστηρίζω. Έχω μία ερώτηση. Στο θέμα της Κροατίας, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την ε, Κροατία και τη Σλοβενία για το ε, θέμα της μεθορίου ή είναι διμερές το ζήτημα αποκλειστικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Σβόμποτα. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος σημείωσε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς με την Τουρκία και συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και συμφωνώ απολύτως. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης Τουρκίας από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος που είναι η Κύπρος. Τι θα γίνει με το πρωτόκολλο της Άγκυρας το Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Επίτροπο για τις εργασίες του. Νομίζω ότι επιτέλεσε πολύ μεγάλο ε, έργο. Σε σχέση με τις θεωρήσεις, ε, συμφωνώ με αυτούς που θεωρούν ότι είναι μεγάλο λάθος να μην συμπεριλάβουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε για τις ε, εργασίες σας κατά την ε, τελευταία εντολή. Σε σχέση με το θέμα των θεωρήσεων, νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι μεγάλο λάθος, επαναλαμβάνει ο μιλητής. Δεν μπορούμε να ζητούμε ε, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μόνο να πληρεί τα κριτήρια. Πρέπει να του βοηθήσουμε. Διαφορετικά ε, ε, δεν θα υπήρχαν πολιτικοί που δεν θα ήθελαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το καθεστώς των θεωρήσεων. Χρειάζεται τεχνική βοήθεια για να υπάρξουν τα νέα βιομετρικά διαβατήρια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια στον τομέα της πρόληψης. Στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα σε σχέση με τη μεθόριο. Η Κροατία έχει ένα πρόβλημα με την ε, Σλοβακία, η Σερβία με το Μαυροβούνιο και ούτω, καθ, ούτω Θα πρέπει να δράσετε προληπτικά έτσι ώστε να μην υπάρχουν γραφειοκρατικά προσκόμματα και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα ως προς το καθεστώς της ε, πρόληψης, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα ως προς τη διεύρυνση. Ο κύριος Κάτσιν έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με τη δήλωσή σας ότι δεν θα πάρετε ένα ειστήριο προς ε, μία ε, κατεύθυνση, μία διαδρομή. Σας χρειαζόμαστε για ακόμα πέντε χρόνια. Αλλά είπατε ότι αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι αρκετά σταθερές. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σταθερές στην αστάθειά τους. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να γίνουν πιο σταθερές και πρέπει να δούμε τι χρειάζεται. Το κοσυφοπέδιο παραγνωρίζεται. Ε, ποιες είναι δυνατότητες ε, για τον, ε, τους Αλβανούς από το Κωσυφοπέδιο να πάρουν θεωρήσεις για να περάσουν στις γειτονικέ χώρες. Πολλοί Αλβανοί έχουν πάει στην Μακεδονία πριν από χρόνια και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ισχυρή πίεση για έκδοση διαβατηρίων στις γειτονικέ χώρες. Αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε κάθε χώρα και ένα καθεστώς απαλλαγής από θεωρήσεις είναι μια από τις προϋποθέσεις και ακόμη μία φράση. Κύριε Επίτροπε, στην Βοσνία έχουμε πολλές κυβερνήσεις, αλλά οι ε, υπουργοί από το επίπεδο της Ομοσπονδίας, της κυβέρνηση κυβέρνησης φεύγουν και έχουμε τώρα μεγάλη κρίση. Πώς μπορούν να πληρώσουν τις ε, τεχνικές προϋποθέσεις χωρίς ε, να τους βοηθήσουμε να έχουν αποτελεσματικές κυβερνήσεις, ζωντανές κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Φλότρετ καμιά εισαγωγή και ίσω μία μόνο ε, ερώτηση, διότι τελειώ μετά από ένα λεπτό θα σα κόψω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω που θα με συγχωρήσετε για αυτή την εισαγωγή, αλλά σοκαρίστηκα διότι δεν άκουσα καμιά αντίδραση από πλευρά σα ε, μετά από τα λόγια ενός συναδέλφου που ήταν Ισλαμόφοβε λόγια και ρατσιστικά λόγια και προσβολές εναντίον του προσκεκλημένου μας. Περιμέναμε λοιπόν από εσά σας κύριε Πρόεδρε μια αντίδραση, μια απάντηση για να κρατήσουμε ε, το κύρος αυτής της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να εμβαθύνετε στην απάντησή σας για την ε, Τουρκία Ήδη μιλήσαμε για τα θετικά σημεία όσον αφορά στην ε, ε, μελλοντική και προσδοκόμενη ε, υπογραφή ενός πρωτοκόλου με την Αρμενία. Υπάρχει μια στρατηγική, ένας τρόπος για την Ευρώπη να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα, την πραγματώση αυτού του πρωτοκόλου. Προς τις μεταναστευτικές ροές η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εδαφικά σύνορα, στα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι η απόκριση της Ευρώπης σήμερα με μια συμφωνία επανεισδοχής δεν είναι η κατάλληλη απάντηση ε, τουλάχιστον για τους ε, μετανάστες και τα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Τι σκέφτεστε να κάνετε ως προς το θέμα αυτό. Ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κροατία. Επίτροπε Ρεν λόγω πρόσφατης εμπειρίας τι συγκεκριμένα βήματα επιμένετε να ληφθούν από την Κροατία για να μην έχουμε το συνεχιζόμενο πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ως προς την Ισλανδία μπορούμε ε, να σκεφτούμε ότι ε, η προσχώρηση της Ισλανδίας θα θέσει τέρμα στα προβλήματα της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Ο κύριος Λάμπστορφ. Κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις για την Τουρκία. Ε, κατά την προηγούμενη θητεία διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα στο θέμα της ελευθεροτυπίας ε, υπήρξαν εντωμεταξύ θετικές ή αρνητικές εξελίξεις. Ε, είπατε ότι στην επόμενη έκθεση πρόοδου θα το εξετάσετε σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα. Δεύτερον, αυτό που είπε η κυρία φλοτρ Χαιρόμαστε για την προσέγγιση Τουρκίας-Αρμενίας αφενός, μια διστακτική προσέγγιση, το ξέρουμε ε, Λίγο πριν έρθετε συζητούσαμε για την ενεργειακή ασφάλεια όμως. Καλό είναι να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια για το ρόλο του Αζερβαϊτζάν στην προσέγγιση Τουρκίας-Αρμενίας, γιατί είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Πώς θα το λύσουμε, ούτω ώστε να υπάρξει μια επικοδομητική κατάσταση, ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Επιτροπέ, μας είπατε τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι πρέπει να κάνει. Τέσσερα πράγματα λέω. Ε, για τις θεωρήσεις, η Βοσνία και το Κωσυφοπέδιο πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική αυτή, γιατί αλλιώς θα αποσταθεροποιηθούν όταν έχει ε, απαλλαγή η Σερβία από τις θεωρήσεις, ενώ αυτές οι δύο χώρες όχι. Δεύτερον, αναγνώριση Κωσυφοπέδιου. Τι θα κάνετε για να πείσετε τις υπόλοιπες χώρες να προβούν σε αυτό το βήμα, ούτως ώστε να λειτουργεί καλά η Ιουλέξ. Ε, τρίτον διαπραγματεύσεις με την Κροατία. Τι κάνετε ε, για τον αποκλεισμό από τη Σλοβενία και Σερβία, μόλις γύρισα από τη Σερβία, τι κάνετε ώστε οι πιστώσεις για την περιφερειακή, διασυνοριακή συνεργασία και τις μειονότητες, ε, γιατί η Βοηβοδίνα για παράδειγμα, να πάνε εκεί στον προορισμό τους και να μην μένουν κολλημένες στο Βελιγράδι όπως φαίνεται ότι συμβαίνει. Ο κύριος Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ρεν και Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο σε μεγάλη πλειοψηφία θα υποστηρίξει την εργασία σας. Δεν ξέρω, πρέπει να αποφασίσετε αν τρέχετε στη Φόρμουλα 1 ή αν είστε μαραθωνοδρόμος. Σχετικά με την Κύπρο είπατε ότι δεν θα αφιστείτε καμιάς προσπάθειας. Τι τεχνικές συμβουλές θα δώσετε για τις διαπραγματεύσεις για την Τουρκία Βεβαίως είναι λεπτό το θέμα. Ποια είναι η μέθοδος και το χρονοδιάγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε ε, για, να, την επισκόπηση του πρωτοκόλου της Άγκυρας και αν ε, θα μεσαλοβήστε ανάμεσα στην Σλοβενία και στην Κροατία για το θέμα που τους απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ με τον κύριο Χάουαρντ κλείνουμε τον δεύτερο γύρο των ε, δέκα παρεμβάσεων και δίνω τον λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω με την Κροατία. Η κυρία Πακ αναφέρθηκε και ο κύριος Πόσελτ και μερικοί άλλοι ομιλητές επίσης και ο κύριος Βόμποντα επίσης. Η έκθεση προόδου θα δημοσιευθεί σε έξι εβδομάδες και συλλέγουμε τα στοιχεία για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να επιφυλαχθώ και θα επανέλθω στην Επιτροπή σας όταν θα έχουμε συμπληρώσει αυτή την εργασία για να σας δώσω πολύ περισσότερο αξιόπιστες εκτιμήσεις ε, για την πρόοδο που έχει γίνει σε ορισμένους κρίσιμους ε, τομείς όπως η δικαστική μεταρρύθμιση και ο τομέας ε, της ναυπήγησης. Πρόκειται για δύο κρίσιμους τομείς και η μεταρρύθμιση παραδείγματος χάρη της δικαστικής εξουσίας έφτασε σε πάρα πολύ λεπτό σημείο και κρίσιμο σημείο και εφαρμόζεται, υλοποιείται και η συμφωνία η οποία επετεύχθη μεταξύ της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Κροατίας για τον τρόπο της εξάλληψης των έξι ναυπηγείων στην Κροατία υλοποιείται και όλα βαίνουν καλώς ως προς τα ναυπηγεία. Αλλά είναι και η μεταρρύθμιση η σημαντική για το άνοιγμα ενός από τους, τα τέσσερα κεφάλαια σχετικά με τον τομέα του ανταγωνισμού και της κρατικής βοήθειας. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό σε μερικές εβδομάδες. Αυτό που μπορώ να πω γενικά είναι ότι η Κροατία έχει κάνει ικανοποιητική πρόοδο για να ανταποκριθεί ε, στα κριτήρια ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά βεβαίως ε, η χώρα υποφέρει, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες υποφέρει από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης και αυτό απαιτεί ε, πολλά μέτρα από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Σχετικά με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως είπα ε, στην εισαγωγή μου, η χώρα κάνει σημαντικές πρόοδους ε, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οκτώ προϋποθέσεις που θέσαμε το Μάρτιο του 2008 και θα αξιολογήσουμε την ετοιμότητα της χώρας, την διαθεσιμότητά της, την δυνατότητα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με βάση τα οκτώ αυτά κριτήρια. Νομίζω ότι υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες η χώρα να το πετύχει αυτό, αλλά και πάλι δεν θα κάνω άλλα σχόλια και θα επανέλθω στην Επιτροπή όταν θα έχω περισσότερα στοιχεία. Αφού παρουσιάσω την έκθεση πρόοδου σχετικά με τη χώρα αυτή. Ο κύριος Βόμποντα έκανε μια ερώτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το διαφορά ανάμεσα στην Κροατία και στην Σλοβενία και ανασχολούμαι με το θέμα αυτό. Εργάστηκα εντατικά επί έξι μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο για το φάκελο αυτό αρχίσαμε από μακριά και πλησιάσαμε. Στο τέλος όμως υπήρξε ανσυμφωνία για μερικές λέξεις και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δυνατότητες ρεαλιστικές να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τα σύνορα. Νομίζω ότι η βοήθεια η συμβουλευτική και η τεχνική ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Τώρα πρέπει οι δύο χώρες και οι ηγέτες τους ε, να προχωρήσουν ακόμα μερικά εκατοστά ε, ως προς την πολιτική τους βούληση για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Η πολιτική ατμόσφαιρα είναι σαφώς πολύ καλύτερη τώρα ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών από ότι ε, στο παρελθόν. Και ενθαρρύνω τους ηγέτες να προχωρήσουν και να βρουν μια διέξοδο για να επιλύσουν αυτό το συνοριακό πρόβλημα και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Φάλερ αναφέρθηκε στη Βοσνία Αρζεγοβίνη και τη βοήθειά μας σχετικά με το θέμα των θεωρήσεων. Είχαμε, παρήχαμε τεχνική βοήθεια στη Βοσνία όπως και σε άλλες χώρες για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ήταν ίσως ε, η πιο ασθενής χώρα ως προς την κεφαλαιοποίηση της ευρωπαϊκής βοήθειας. πολλά από τις χώρες μέλη ε, που έχουν δώσει ε, γνώσεις, συμβουλές, ε, διευκολύνουν αυτή την απελευθέρωση με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Δεν πρόκειται μόνο για μια πολιτική απόφαση. Απαιτεί πολύ τεχνική εργασία, η οποία καμιά φορά είναι πολύ βαρετή, αλλά είναι απαραίτητη. Ο κύριος Κάτσιν αναφέρθηκε στη σταθερότητα της αστάθειας της περιοχής και πάλι καταλαβαίνω μέχρι ενό ορισμένου σημείου, αλλά από την άλλη πλευρά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ε, μια ε, σταθερή αλλά αργή διαδικασία σταθεροποίηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Και ελπίζω ότι η κατάσταση αυτή και η εξέλιξη αυτή θα ε, συνεχιστεί και θα αποδώσει περαιτέρω αποτελέσματα. Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά στα προβλήματα της διακυβέρνησης στη Βοσνία ε, τα οποία αναφέρθηκαν μέσα από τον κύριο Τάλερ. Είναι σαφές ότι έτσι όσο έχει η κατάσταση στη χώρα τώρα, η Βοσνία Αρζεγοβίνη δεν είναι έτοιμη ε, για ε, αρχίσει διαπραγματεύσεις ενταξιακές. Δεν έχουμε ένα ε, μανιφέστο, αν θέλετε, για την μεταρρύθμιση στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχουμε δύο βασικές ε, προϋποθέσεις. Είναι η μία ότι η χώρα θα μπορεί να μιλάει με μία φωνή όταν θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια χώρα να μπλοκάρει την λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της διέρεσης της χώρας, των πολιτικών δυνάμεων. Και δεύτερον, θέλουμε να έχουμε ε, πιο αποτελεσματική κρατική δομή, ούτω ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις υποχρεώσεις της προενταξιακής διαδικασίας. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι όταν επιτευχθεί η μετάβαση από ε, μια, από τον ε, ανώτατο εκπρόσωπο προς ε, μια ενισχυμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί η Βοσνία Ερζεγοβίνη να ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις και θα είναι μεγάλη πρόοδος για τη χώρα και θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία πολιτική για μια μεταρρύθμιση συνταγματική. Αυτό το βλέπω περισσότερο ως εξέλιξη και όχι ως επανάσταση ως προς το Σύνταγμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ας εστιαστούμε στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, διότι είναι μια από τις χώρες κλειδί στα Δυτικά Βαλκάνια, σημαντικότατη και ελπίζω ότι τον Οκτώβριο το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με την Βοσνία Ζεγοβίνη. Βεβαίω η Προεδρία θα πρέπει, είναι ευθύνη τη Προεδρία και θα, ε, το Συμβούλιο θα μπορούσε να λάβει χώρα τον Νοέμβριο ότως ε, ούτως ώστε να περάσουμε, να έχουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο και να έχουμε μια ενισχυμένη παρουσία. Αναφέρθηκε η Τουρκία και η πρόοδος, η έλλειψη πρόοδου. Και πάλι θα ήθελα να αναφερθώ στο πακέτο διεύρυνσης και στην έκθεση πρόοδου που θα παρουσιαστεί σε μερικές εβδομάδες και τότε θα έχουμε μια πιο ε, σταθερή ανάλυση και πιο αντικειμενική αξιολόγηση τότε. Υπάρχουν δύο ή μάλλον τρία σημαντικά θέματα που εξελίσσονται στην Τουρκία. Πρώτον είναι η πρωτοβουλία η κουρδική. Πρέπει να δούμε αν η κυβέρνηση της Τουρκίας και το κοινοβούλιο θα μπορέσουν να ενισχύσουν μια σοβαρή πρωτοβουλία ούτως ώστε στη νότια-ανατολική πλευρά της χώρας να εξελιχθεί η κατάσταση με τους Κούρδους. Δεύτερον, οι σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας. Υπάρχουν θετικά σημεία, παραδείγματος χάρη χτες. Και τρίτον, το πρωτόκολλο της Άγκυρας, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις η Τουρκία που απορρέουν από το πρωτόκολλο αυτό. Ο κύριος Λάμπστορ έθεσε το θέμα σχετικά με το ρόλο του Αζερβαϊτζάν μέσα στο πλαίσιο αυτό της ενεργειακής ασφάλειας, των σχέσεων με την Αρμενία κλπ. Πρόκειται για μια εύστοχο ερώτημα και εν συντομία φαίνεται ότι γενικά η διαμάχη του Ναγκόρνο καραμπαχ παρεμποδίζει την έναρξη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Αρμενία ε, και έχει και κάποια σχέση με την, ε, τις ενεργειακές προμήθειες από το Αζερβαϊτζάν. Νομίζω ότι ε, επιτελείται κάποια πρόοδος και μπορούμε όλοι να υποστηρίξουμε αυτή την τάση και όπως είπα προηγουμένως, όταν η Τουρκία και η Αρμενία μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις τους, να έχουν διπλωματικές σχέσεις, θα έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα που θα είναι πάρα πολύ θετικό για την σταθερότητα και την πρόοδο στην περιοχή του Καυκάσου. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Α, υπήρχε άλλη μία ερώτηση, με συγχωρείτε. You uh, ε, ήταν τόσες οι ερωτήσεις, ναι, κατανοώ ότι ήταν, ε, είναι οι δυσκολότεροι. Τι πιστεύετε για την Ιούλεξ και την ε, Σερβία ως προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Αληθεύει, υπάρχει μία κίνηση στη χώρα που αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο. Ποια είναι η απόψή σας στην Σερβία ή στο Κωσυφοπαίδιο. Εκτός μικροφώνου η απάντηση. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Γιούλεξ ε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο έτσι ώστε να υπάρξει έλεγχος της μεθορίου με το κοσυφοπέδιο και είναι ύψης της σημασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην ε, περιοχή αυτή. Άρα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των ε, οριοθετήσεων που έχουμε θέσει μέσα στα πλαίσια του οδικού χάρτη και αυτό τονίστηκε και στην έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σε σχέση με την ανταπόκριση των ε, προαπαιτήσεων, των benchmarks. Βεβαίως, αφού προτείναμε την συνεργασία με την EULEX προς τη Σερβία, η Σερβία δέχτηκε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα προσκόμματα από πλευράς κοσυφοπεδίου, αλλά θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Όπως ξέρετε, πρόκειται για, πρόκειται για προνόμιο του Συμβουλίου και ο Χαβιέ Σολάνα και ο Πίτερ Φέιθ είναι αυτοί που βρίσκονται στην ε, πρώτη ε, γραμμή για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο τελευταίος γύρος περιορίζεται σε 30 δευτερόλεπτα. Θα σας αφαιρέσω το λόγο, εάν υπερβείτε τα 30 δευτερόλεπτα. Λαντσμπέργκης. Uh, Ευχαριστώ. Επίτροπε. Χτες μόλις ε, άκουσα για το θέμα των περαιτέρω διευρύσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που έχουν γενικές, ε, γενικότερες αντιρρήσεις Άρα θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα λάβει χώρα η διεύρυνση και ποια θα είναι η πραγματική μας θέση. Πώς θα αντικαταστήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης. Μήπως θα έπρεπε να μπούμε σε μία περίοδο περίσκεψης σε σχέση με την διεύρυνση. το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα θέματα που αφορούν την Τουρκία εν ώψη της αξιολόγησής της. Πρώτον, ο συνεχιζόμενος επικισμός της Κύπρου, ο αριθμός των επίκων σήμερα υπολογίζεται γύρω στο μισό εκατομμύριο σε ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Και δεύτερον, η τουρκική κατοχική στρατιωτική παρουσία η Κύπρος είναι η πιο στρατικοποιημένη περιοχή στον κόσμο και ακόμα χθε ο τουρκικός στρατός δεν επέτρεψε, δεν επέτρεψε σε προσκυνητές να προσκυνήσουν σε εκκλησία στα κατεχόμενα. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει σε δύο αυτά μεγάλα θέματα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια, διότι από ό,τι κατανοώ πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία και κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχει αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να συνεχίσετε να εργαζόσαστε με τον κύριο, να συνεργαζόσαστε με τον κύριο Καρλ Μπίλντ και ο στόχος σας, το δικό σας σχέδιο είναι το μόνο ρεαλιστικό, η μόνη ρεαλιστική βάση για να εξεύρουμε μία λύση, για να υπάρξει μία καλύτερη ατμόσφαιρα. Τάραντ. Ορισμένες από τις απαντήσεις σας ε, έχουν δώσει απάντηση. Απλώς ε, για να τονίσω κάτι, Θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία να λήξουν το 2010 ή θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο υπομονετικοί. Ονορεύολε Θα εγγραφώ την επόμενη φορά πρώτος, για να μην έχω αυτούς τους περιορισμούς. Ένα, μια πολιτική σκέψη. Έχουμε την ε, εντύπωση ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει απαγκιστρωθεί από τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρώπης και από το θέμα της ε, θεσμικής σταθερότητας της Ευρώπης. Υπάρχει εξής ανησυχία. Εάν δεν υπάρχει ένα κοινό εγχείρημα, τότε η διαδικασία δεν θα έρθει σε αίσιο πέρας. Θα πρέπει να ε, ίσως να προφούμε σε μια διαδικασία περισυλλογής. Κουμουτσάκος. Η χώρα μου στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στην λογική της πλήρου συμμόρφωσης για την πλήρη ένταξη. Full compliance, full membership. Η Τουρκία όμως απέχει πάρα πολύ από το full compliance, άρα απέχει πάρα πολύ και από το full membership. Η Ένωση οφείλει να διαφυλάξει την αξιοπιστία της όταν βλέπει ότι οι δεσμεύσει και υποχρεώσει κρατών, υποψηφίων κρατών απροκάλυπτα δεν τηρούνται. Θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογε συνέπειε και κυρώσει. Κύριε Επίτροπε, είσαστε στο στάδιο σύνταξης της έκθεσης προόδου της Τουρκίας που θα παρουσιάσετε τον Οκτώβριο. Θα παρακαλούσαμε και νομίζω ότι επιβάλλεται να είναι μια έκθεση που θα καταγράφει με ακρίβεια και χωρίς ερωποιήσει την τακτική αυτής τη Τουρκίας να μην ανταποκρίνει τι υποχρεώσει της. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία σας για το θέμα των θεωρήσεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά νομίζω ότι οι ενδείξεις μας δείχνουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα πρωτόκολλο με την Σερβία, ούτως ώστε η Σερβία να μην εκδίδει σερβικά διαβατήρια στα, στους κατοίκους της, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και πώς ε, θα επιτύχουμε η Σερβία να μην υπονομεύει ε, την Σερβία η Σνογοβίνη ε, και θα εξασφαλίσει τα σύνορα και πώς η Σερβία θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν τον οδικό χάρτη αν δεν παραδώσει τον Μλάντιτς. Εάν δεν υπάρχει δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ο κύριος Πρέβριτς. Είπατε ότι έχει γίνει μία προσπάθεια και πρόοδο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε τον άκρατο εθνικισμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση των Σκοπίων σε βάρος της Ελλάδας. Σας έχω εδώ μία φωτογραφία όπου ο Πρωθυπουργό ε, του κράτους των Σκοπίων καταθέτει στεφάνι στο υποτιθέμενο μνημείο της Μεγάλης Μακεδονίας όπου ζητείται υποδούλωση της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του βόρειου τμήμα της Ελλάδος. Πώς μια τέτοια χώρα που ε, είναι επιθετική σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ε, έχει ενταξιακή πορεία. Δεύτερον, δύο δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της Τουρκίας. Θέλετε Σόνι και καλά να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα που το μέρο μέρος είναι στην Ασία. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε, ο κύριος Ρεν μίλησε για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Τουρκία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και δεσμεύσεις απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Είπαμε ότι η Τουρκία πρέπει να τηρήσει όλους τους όρους και ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συμβαδίζει με τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Αυτό δεν γίνεται. Εξακολουθούμε να ανοίγουμε νέα κεφάλαια, ενώ τίποτα δεν συμβαίνει στην Τουρκία. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατικό, ο Ευρωπαίος, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν μας ακολουθούν πια, πόσα, ε, τι θα κάνουμε για αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, πώς η Τουρκία θα μπορέσει να τηρήσει τους όρους και να πληρεί τα κριτήρια. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ αισιόδοξο. Αυτό δεν είναι μια κριτική, διότι όταν είναι κανεί αισιόδοξο ζει καλύτερα. Μια γενική ερώτηση. Η διαδικασία διεύρυνση ε, με βάση την, ε, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Τι σκέφτεστε γι' αυτό. Φτάσαμε στο τέλος της ε, συζήτησης και ο Επίτροπος έχει το λόγο για την, τις τελικές απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ακούσαμε πολύ σοβαρά πράγματα να τίθενται ο κύριος Λαντσμπέργκης πρώτος μίλησε για εναλλακτικέ στην διεύρυνση. Εμείς τώρα θέλουμε να κάνουμε μια ε, ε, σταθεροποίηση, παγίωση του, των εξελίξεων των προηγουμένων ετών και ε, τώρα υπάρχει μετά από την, ε, τις προηγούμενες διευρύνσεις πρέπει να δούμε ότι θα υπάρξει και μια φάση παγίωσης ε, των 27. Σε σχέση με τις υφιστάμενες ε, υποχρεώσεις στον τομέα της διεύρυνσης μπορώ να αναφέρω μόνο την, την επανειλημμένη συνένεση που είχαμε το Δεκέμβριο του 2006 μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν και ισότιμη αφορά προσυπογράφω τη συνένεση αυτή. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη ε, προοπτική για να πετύχουμε τους στόχους μας σταθεροποίησης και ολοκλήρωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ας ε, εμείνουμε στις υφιστάμενες υποχρεώσεις δεσμεύσεις μας, χωρίς να προσθέσουμε άλλες δεσμεύσεις στον τομέα της διεύρυνσης. Ας ε, μείνουμε στις χώρες που έχουν ήδη την ευρωπαϊκή προοπτική. Κατόπιν τούτου, η ε, εταιρική σχέση στην Ανατολική Ευρώπη είναι μεγάλη θεσμική βελτίωση, μεγάλη πρόοδος, ε, ένα ε, εγχείρημα που εξελίσσεται ακόμη και στην πορεία της εφαρμογής έχουμε μια διαδικασία εκμάθησης. Η εταιρική σχέση είναι σημαντική ε, για πολλούς λόγους, γιατί περιλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να γίνει για να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και χωρών της ανατολικής διάστασης. Θα πρέπει να κεφαλοποιήσουμε την, τις, τις πρωτοβουλίες αυτές για τη βελτίωση των σχέσεων και με την Ουκρανία και με τις άλλες χώρες της περιοχής ο κύριος Μαυρονικόλας και ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Πλεύρης ε, και οι τρεις αναφέρθηκαν στην Κύπρο και την Τουρκία. Εγώ έχω απαντήσει ήδη στις ερωτήσεις αυτές και προσθέτω μόνο ότι στην έκθεση πρόοδου για την Τουρκία θα αναλύουμε και την πρόοδο αλλά και τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται ε, στην ε, Τουρκία όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Και μετά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα συναγάγουν συμπεράσματα με βάση τις συστάσεις της Κομισιόν. Είναι προφανές ότι η Τουρκία υποχρεούται να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας και σε σχέση με την Κύπρο και την Τουρκία είναι τεράστια σημασία να συμβάλλει η Τουρκία προς, μια ένα ευνοϊκό πολιτικό κλίμα και σοβαρές συνομιλίες ε, για την επίλυση του Κυπριακού. Ο κύριος Βάιγκελ μίλησε για το θέμα αυτό των συνορων κροατια Κροατίας-Σλοβενία, συνέχιση διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Θα πρέπει βεβαίως να ε, φτάσει η ενθάρρυνση αυτή μέχρι τους ηγέτες των δύο, των δύο χωρών και αν χρειαστεί θα ε, διαβουλευτούμε μαζί σας. Ο κύριος Τάραντ έθεσε το θέμα της Ισλανδίας και αν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις το 2010 ή αν θα πρέπει να ε, κάνουμε υπομονή. Η πολιτική μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Προτιμούμε την ποιότητα σε σχέση με την ταχύτητα και γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας γιατί οι πρώτες σοβαρές ενδείξεις της ετοιμότητας της Ισλανδίας να, να πληρώσει τις ε, προϋποθέσεις ε, ε, θα γίνουν όταν ετοιμαστεί η γνωμοδότηση για την χώρα αυτή. Ο κύριος Βανόρντεν στο προηγούμενο γύρο έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αν η προσχώρηση της Ισλανδίας θα οδηγήσει στο τέλος της κοινή πολιτικής αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι και στη, όταν μιλάμε για την Ισλανδία και οποιαδήποτε άλλη χώρα, η Ισλανδία ε, είναι εκείνη που θα πρέπει να προσαρμοστεί στο κοινοτικό κεκτημένο. Δεν θα γίνει το αντίστροφο και η ίδια αρχή ισχύει και για την Ισλανδία όπως και για την Τουρκία και οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα ή ενδεχομένως ε, πιθανή η χώρα. Ο κύριο Πανσέρη μίλησε για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη. Τα γνωρίζω όλα αυτά και νιώθω την αγωνία των πολιτών μα. Ευτυχώ ε, υπάρχουν κάποια δείγματα ανάκαμψη και το σχέδιο οικονομική ανάκαμψη. εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί μπορέσαμε να αποφύγουμε τη βαθιά και μακρά οικονομική ε, κρίση ε, βέβαια η διεύρυνση δεν είναι ο λόγος των οικονομικών μας προβλημάτων. Η δημοσιονομική, οικονομική κρίση και η ύφεση δεν ε, ε, άρχισαν στην Πράγα ή το Βελιγράδι, αλλά στη Wall Street και προκλήθηκαν από συστημικά λάθη του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Αυτά θα πρέπει να διορθωθούν η διεύρυνση δεν πρέπει να καταστεί από διοπομπαίος τράγος και να φορτωθεί ε, λάθη που δεν προκάλεσε. Η Βαρόνι Λάντφορντ μίλησε για ένα πιθανό πρωτόκολλο με τη Σερβία για την έκδοση ή μη έκδοση διαβατηρίων προς τους, ε, για τους ε, κατοίκους της Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Αυτό το ξέρουμε δεν είναι πρόβλημα ακόμα, γιατί αν ε, δεν περάσει πολύς χρόνος μέχρι την απαλλαγή των θεωρήσεων, δεν θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, τα καθεστώτα που αφορούν τις, χωρί... τις ε, θεωρήσεις ε, ως γενικό κανόνα βασίζονται στην αρχή της ιθαγένειας και η Σερβία έχει ακολουθεί συγκεκριμένη πρακτική σε αυτό το τομέα και από εκεί απορρέουν και κάποια δικαιώματα. Στην πράξη όμως δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή δεν προβλέπω ε, να παίρνουν πολλά διαβατήρια οι κάτοικοι τη Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Και βεβαίως το έχουμε συζητήσει αυτό και με τους ηγέτες τη Σερβίας. Ο κύριος Κούκαν αναφέρθηκε σε κάποια θέματα που δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω. Περιορίζομαι να πω, για να απαντήσω και στον παλιό φίλο, τον κύριο Κούκαν και τον κύριο Παντσέρη, Λέω ότι οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου, άρα είναι πολύ σημαντικά και για τις διαπραγματεύσεις ε, διεύρυνσης. Η διαδικασία ένταξης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στηρίζεται πιο πολύ στην εσωτερική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι ενδιαφερόμενες χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους ευρωπαϊκούς ε, νόμους ε, κανονισμούς που με τη σειρά τους έχουν οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τέλος, ε, και αυτό είναι καλό για να τελειώσουμε, αναφερόμενο στον κύριο Κούκαν ακόμη, ως ο Επίτροπος για τη διεύρυνση εξορισμού πρέπει να είναι επαγγελματίας αισιόδοξο ε, και θα συνεχίσω και στις, ε, στα πλαίσια της συνεργασίας μου μαζί, σας να είμαι αισιόδοξο. Ευχαριστούμε όλοι τον Επίτροπο για την εισήγησή του, για τις απαντήσεις, τις ανταπαντήσεις. Ε, θα ξαναβρεθούμε στις 3 η ώρα. Μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα και μετά τις ψηφοφορίες όπως προβλεπόταν χτες θα έχουμε μία συνάντηση με τον δόκτορα Μόρα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Τέλος, σας ζητώ συγνώμη διότι χρειάστηκε να σας διακόψω, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή για να τηρήσουμε το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα τα πούμε στις 3.